Thank you, colleagues. If you can please take your seats. We... Καλημέρα, συνάδελφοι. I still see colleagues um, uh, greeting each other, please take your seats. Thank you. So, colleagues, um, uh, happy new year to all of you. Πρώτα απ' όλα να σας ευχηθώ, αγαπητοί συνάδελφοι, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, λοιπόν, σε όλους σας. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με κοινή συζήτηση και αν συμφωνείτε με αυτό το τμήμα της ημερησίας διατάξεως θεωρείται εγκεκριμένο. Έχουμε και ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να έχετε όλοι έτοιμες ε, τις ε, ε, κάρτες ψηφοφορίας και αν δεν τις έχετε να σας τις φέρουν. Φτάνουμε λοιπόν εδώ και στρέφομαι προς την κυρία Γκρέσλερ η οποία είναι η συμπρόεδρος από την Επιτροπή με την οποία θα συνεργαστούμε σήμερα έτσι ώστε να συζητήσουμε τα θέματα της καταπολέμησης της απάτης. Θα δώσω τον λόγο στην συμπρόεδρο καθώς επίσης και στον κύριο Λόπες Αγγιλάρα, τον εισηγητή. Πριν ξεκινήσουμε βέβαια θα ήθελα να πω και δύο λόγια σχετικά με την σημασία του συμφωνηθέντος κειμένου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Από, άποψη, από την άποψη της ΛΥΜΠΕ χαίρομαι που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Κύριε Γκρέσλ, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους και καλή χρονιά. Αυτό ισχύει και για την ε, δική μας επιτροπή, αυτό που είπατε για την επιτροπή του ελέγχου του προϋπολογισμού. Είναι ε, ιστορική ας πούμε μέρα σήμερα, είναι πολύ σημαντικό ε, αυτό το οποίο έχουμε επιτύχει και είναι κάτι το οποίο επιτύχαμε μέσω πολύ σκληρής εργασίας κατά τη διάρκεια των διακοπών και με τον τρόπο αυτό καταφέραμε να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Ε, είναι σημαντικό επίσης που συζητούμε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και είναι σημαντικό να δούμε την οδηγία αυτή ε, η οποία θα πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε ευθυγράμμιση και εναρμόνιση έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν οι διάφορες διατάξεις του ποινικού δικαίου. Δουλέψαμε 4,5 χρόνια ε, γιατί ξεκινήσαμε την εργασία το καλοκαίρι του 2012 και ε, ε, αυτή η εργασία αποτέλεσε βάση και για την ε, εισαγγελία, η οποία θα πρέπει να έχει αρμοδιότητες σχεδόν αποκλειστικές επί του θέματος. Θα ήθελα μόνο να πω σήμερα ότι αν επιδιώξουμε να συμφωνήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε και το Συμβούλιο και ξέρουμε πόσο δύσκολα μπορεί να είναι τα πράγματα με το Συμβούλιο. Λόπε Αγγιλάρ ε, θα, νομίζω θα συμφωνήσει μαζί μου. Νομίζω θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Σλοβενική Προεδρία ε, και κύριε Κοντλάρη και Χρόσικ, ε, σας ευχαριστούμε για όσα κάνατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης ε, την Ιταλική, τη Λετωνική και την Ολλανδική Προεδρία για την επίτευξη των στόχων και Υπάρχουν διάφοροι υπάλληλοι κρυμμένοι στο Συμβούλιο, οι οποίοι εργάζονται πάρα πολύ αποτελεσματικά και θα πρέπει ο Λορένσο Ματέο, ο Λορένσο Σαλαζάρ ε, να λάβουν τις ευχαριστίες μας. Ε, Μάρζο Ριμπόν και Νίκορας Φράντζεν από την Ολλανδική Προεδρία, παραδείγματο χάρη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά αυτού του υπαλλήλου γιατί είναι ιστορικό το σημερινό επίτευγμα ε, είναι ορόσημο διότι μέχρι στιγμής ε, δεν είχε εξευρωπαϊστεί ούτως επίνο ο τομέας. Η κυρία Σρέντερ, η κυρία Όλριχ, Χόφμαν, Νικολάη, ε, Γιόνκερ, όλοι αυτοί οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να λάβουν επίσης ευχαριστίες μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους γλωσσομαθείς νομικούς. Σήμερα κατορθώσαμε να συμφωνήσουμε για ένα ιδιαίτερα σημαντικό συμβαστικό κείμενο. Ε, συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ ήταν οι ενό σε 10 εκατομμύρια και δύο ε, τουλάχιστον κράτη-μέλη πλήττονται, οπότε νομίζω ότι για τη δυσυναριακή συνεργασία είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς που τελικά καταφέραμε να συμπεριληφθεί μέσα στο κείμενο. Έχουμε το άρθρο 18 για το όριο. Κατορθώσαμε να εγκριθεί αυτή η διάταξη. Ε, και φυσικά θέλουμε να αποφύγουμε ένταση της εγγραφειοκρατίας. Ε, στο άρθρο 5 επίσης ε, έχουμε μεγάλη επιτυχία διότι έχουμε τα ελάχιστα όρια, τις ελάχιστες ποινές. Τέσσερα χρόνια, 100.000 ευρώ εγκρίθηκε αυτό στο Συμβούλιο και επίσης ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό ισχύει για, όλα τα, για όλες τις αξιόπινες πράξεις, για όλα τα κράτη-μέλη. Μιλήσαμε και για την εφαρμογή των δικαστικών υποθέσεων, για την παραγραφή. Ε, και ε, είχαμε ζητήσει 8 χρόνια και θα δούμε, διότι τελικά εγκρίθηκε στη διάταξη για την αναθεώρηση. Ε, πρόκειται για συμφωνία σε πρόορη δεύτερη ανάγνωση και αν συμφωνήσετε θα γράψουμε μια επιστολή προς το Συμβούλιο όπου θα αναφέρουμε ότι χωρίς τροπολογίες συμφωνεί και το Κοινοβούλιο εάν τελικά εγκρίνει και τις κατευθυντηρίες γραμμές στο τελικό σχέδιο το Συμβούλιο. Είναι ιστορική στιγμή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και ελπίζω να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία, αλλά πριν θα ήθελα να ζητήσω τον κύριο Λόπελ Αγγιλάρο, ο οποίος ε, είναι εισηγητής να πει δύο λόγια. Ναι, και εγώ θα ήθελα να, δράξω να την ευκαιρία έτσι ώστε να ευχηθώ καλό 2017 σε όλους. Βεβαίως προσυπογράφω κάθε μία από τις λέξεις και τα λόγια τα οποία ε, είπατε εσείς ο ίδιος και η κυρία Γκρέσλερ. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της οδηγίας PIF ε, και είναι σημαντικό να προωθηθεί γιατί ήταν πραγματικά ένας από τους πιο περίπλοκους φακέλους που εκλήθημε να αντιμετωπίσουμε. Ε, είναι ε, μεγάλη η ιστορία η οποία έχει ξεκινήσει ε, και το ποινικό δίκαιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η χρήση του δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντιμετώπισε καχυποψία, δυσκολίες και κυρίως σε σχέση και με την συμπερίληψη του ΦΠΑ στις Στου ίδιου ε, πόρου, ε, γιατί ο ΦΠΑ είναι πραγματικά ένας ε, ευρωπαϊκός ο πόρος, ίδιος πόρος και νομίζω ότι με την ίδια ζέση και εμεί προσπαθήσαμε να δουλέψουμε έτσι ώστε να εγκριθεί αυτή το, η, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το κείμενο βεβαίως δεν είναι τέλειο, ε, είναι αποτέλεσμα συμβιβασμών και δίνει την ε, δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ε, οι βάσεις του ποινικού δικαίου έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να φτάσουμε ε, χρόνο σε την ε, εισαγγελία. Οι διαδικασίες βρίσκονται σε πολύ ε, δύσκολη φάση. Εμείς προετοιμάζουμε τα πράγματα έτσι ώστε ομαλώς να οδηγηθούμε ε, προς αυτήν την ολοκλήρωση. Χρειάζεται ακόμα προσπάθεια, χρειάζονται πρόοδοι, αλλά το κείμενο πιστεύω ότι είναι ισορροπημένο. Συμπεριλαμβάνει την απάτη ΦΠΑ, την δυνατότητα οι απάτες δημοσίων προμηθειών να αναφερθούν ε, και να συμπεριληφθούν εις ε, την ενδιάμεση αξιολόγηση στην, ε, εντός της διετίας με ελάχιστες περιόδους όσον αφορά την παραγραφή και όσον αφορά τα όρια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω βεβαίως τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις ε, τους υπαλλήλους, ε, την γραμματεία, ε, βεβαίως την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, την κυρία Γκρέσλε προσωπικά και όλους εσάς αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν στην διαδικασία και από τις δύο επιτροπές. Σας περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία, στο κείμενο στο οποίο έχουμε συμφωνήσει. Άρχεται η ψηφοφορία. Has everyone voted? Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Και εγκρίνεται 47 υπέρ, 8 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια σε όλους. So colleagues, uh, Mrs. and I will now... Κύριε Γκρέσλη και εγώ θα στείλουμε τώρα μια επιστολή στην ε, Μαλτέζικη ε, Προεδρία, όπου αναφέρεται ότι αν το Συμβούλιο εγκρίνει το κείμενο ε, και εμεί ε, θα συστήσουμε να ψηφιστεί χωρί κάποια τροποποίηση σε δεύτερη ανάγνωση το κείμενο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκρέσλε. Ενώ αποχωρούν οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, α ε, υιοθετήσουμε την ημέρα διάταξη τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Περνώ στο σημείο 2, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Σα παρακαλώ να κάνετε ησυχία καθώ αποχωρούν οι συνάδελφοι. Έχουμε και μερικέ ανακοινώσει. Κύριε Γκάμπριελ, δικαστικό. Συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά υποτίθεται ότι θα υπήρχε και μια δεύτερη ψηφοφορία για τις θεωρήσεις ε, της Γεωργίας. Yes, we're coming to Ναι, θα φτάσουμε και εκεί, μην ανησυχείτε. Uh, Είναι στο σημείο 5 της μέσης διάταξης της δικής μας. Μην ανησυχείτε, δεν το έχουμε ξεχάσει. We're just going to make some uh, chairs announcements and then we'll reach the vote. Don't worry. Πρώτα θα κάνουμε κάποιες ανακοινώσεις και μετά θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Μην ανησυχείτε. Συνάδελφοι, ησυχία, γιατί έχω αρκετές ε, ανακοινώσεις, μία όμως ε, είναι πιο σημαντική. Παρακαλώ ποιος θέλει να αποχωρήσει να το κάνει ήσυχα. Ευχαριστώ. Συναδελφοί, πρώτη η ανακοίνωση του Προέδρου. Εφόσον είναι η πρώτη συνεδρίαση μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Βερολίνο στις 19 Δεκεμβρίου, θα θυμάστε και εσείς συνάδελφοι ότι έλαβαν χώρα στο Βερολίνο λοιπόν αυτές οι επιθέσεις. 12 ε, άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πάνω από 40 τραυματίστηκα. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να πατήσω φόρο τιμής ε, στα θύματα, στις οικογένειές τους, Γερμανού Γερμανούς πολίτες ε, εν γέννη και στις ε, γερμανικές αρχές. Ξέρετε ότι παραδοσιακά και στην Επιτροπή μας εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας όταν ε, σημαίνουν τέτοια γεγονότα και αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Θα ήθελα να ε, διαβεβαιώσω τους Γερμανούς συναδέλφους ε, της Επιτροπής μας ότι είμαστε πραγματικά αλληλέγγυοι μαζί τους ε, και να τους εκφράσουμε τα θερμά, τους, θερμά μας συλληπιτήρια και σας παρακαλώ τώρα να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης. you very much. Colleagues, our, our uh, other announcements. Uh... Συνάδελφοι, να περάσουμε στις επόμενες ε, ανακοινώσεις ε, για τους συζητητές. Κυρία Γραπίνη, από τους σοσιαλιστές για την πρόταση της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της ανταλλαγής ε, αυτοματοποιημένων δεδομένων σε ό,τι αφορά την καταχώρηση για ταξινόμηση ε, οχημάτων στην Δανία. Ο κ. Φοντάνα ε, είναι εισηγητής για τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες και τα σχετικά μέτρα ελέγχου. Συμφωνεί η Επιτροπή. Ναι. Και τώρα, σε ό,τι αφορά τις της πράξης. Στην συνεδρίαση τη 14 η Νοεμβρίου, οι συντονιστέ συμφώνησαν να παρατείνουν ε, την προθεσμία για, τις, ε, για την υποβολή αντιρρήσεων μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Σε ό,τι αφορά τον ε, κανονισμό της 3ης Οκτωβρίου για το κοινό πλαίσιο παρακολούθηση αξιολόγηση, για τον κανονισμό 514 του 14 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που θεσπίζει γενικές διατάξεις για το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και σε ό,τι αφορά την ε, αστυνομική συνεργασία κτλ. Θα ήθελα να συνημερώσω ότι δεν έχουμε λάβει ενστάσεις και τέλος ε, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ στις 8 Δεκεμβρίου είχαμε τρεις κατεξιώσεις πράξεις ε, που συμπληρώνουν τα παραρτήματα του κανονισμού 98 13 σε ό,τι αφορά τις πρόδρομες εκρηκτικές ύλες. Είχαμε την προθεσμία τη 14 η Δεκεμβρίου για την υποβολή ενστάσεων, αλλά δεν υπήρξαν. Και τέλος, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 15-16 Φεβρουαρίου, 8 Σεπτεμβρίου και 10 Οκτωβρίου του 2016. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, εγκρίνονται. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για, την, ε, για το 2017, ε, ηλεκτρονική ψηφορία για τις τρίτες χώρες υπήκο των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση θεώρηση για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των ε, κρατών μελών και πιο συγκεκριμένα για τη γεωργία. Οι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι υπήρξε συμφωνία στον, στον τελευταίο τριμερή διάλογο στις 13 Δεκεμβρίου ε, και στις 20 Δεκεμβρίου είχαμε και επιβεβαίωση από την Κορεπέρ. Θα ψηφίσουμε τώρα, όμως να δώσουμε το λόγο στην κυρία Καμπριέλα αν θέλει ε, να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο μηνύματα έχω. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως όλους τους συναδέλφους των πολιτικών ομάδων για την ε, υποστήριξη, γιατί από την αρχή συμφωνήσαμε όλοι ότι η Γεωργία καλύπτει πλέον όλες τις προϋποθέσεις και επομένως θα πρέπει ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει αυτό το τελευταίο βήμα έτσι ώστε οι γεωργιανοί πολίτες να μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα δεύτερο μήνυμα προς το Συμβούλιο έτσι ώστε να ολοκληρώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα τις εσωτερικές τεχνικές διαδικασίες έτσι ώστε στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στέλνοντας ταυτοχρόνως ένα καθαρό μήνυμα σε όλους τους πολίτες της Γεωργίας. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ κυρία Γκαμπριέλ. Ε, αυτά τα μηνύματα είναι σαφή ε, όσον αφορά αυτό το θέμα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θέλει κάποιος άλλος το λόγο και επομένως μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία επί του συμφωνημένου κειμένου. Άρχεται η ψηφοφορία. Colleagues, if I could um, just ask for the EPP to Υπάρχει ένα προβληματάκι με το ΕΛΚ, υπάρχουν δύο παραπάνω ψήφοι. Ε, φαίνεται ότι ξεκινήσε το ΕΛΚ ενθουσιοδός την νέα χρονιά. Τώρα έχουμε έναν επιπλέον ΕΛΚ. Still one, if, one could just um, opt out. I know everyone wants to vote on this. Ωραία. Να να είμαστε σωστοί στον αριθμό. Ξέρω ότι όλοι θέλετε να ψηφίσουμε. Έφυγε και ο τελευταίος επιπλέον ΕΛΚΑ. Ωραία. Ε, ψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία εγκρίνεται 45 ψήφοι υπέρ, ε, συγγνώμη, 42 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Σημείο 6, παρουσίαση των προτεραιοτήτων ε, της ε, Προεδρίας ε, της Μάλτας. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Αντέλα που είναι Υπουργός ε, Εσωτερικών Υποθέσεων, τον κύριο Μπονίτσι, ε, Υπουργό Δικαιοσύνης και Πολιτισμού. Ε, σας καλωσορίζω και τους δύο και βεβαίως εύχομαι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα εις την διάρκεια της Προεδρίας σας. Χαίρομαι που είστε εδώ Ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, γι' αυτό θέλω να ξεκινήσουμε έγκαιρα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνετε και οι δύο από μία σύντομη ε, εισήγηση ε, και μετά τα διάφορα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα υποβάλουν τις ερωτήσεις τους. Ξέρετε ότι αυτή είναι η συνήθις διαδικασία η οποία σας έχει γνωστοποιηθεί. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην μακρηγορήσετε ιδιαιτέρως έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Σας καλωσορίζω για μια ακόμα φορά θερμότατα. Ε, κύριε Αμπέλα, μπορεί να ξεκινήσετε εσείς με την δική σας δήλωση πρώτα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. είμαι ευτυχής που μπορώ να παρουσιάσω ενώπιόν σας τις προτεραιότητες ε, της ε, ε, Μαλτέζικης Προεδρίας. Τα τελευταία έξι χρόνια η Ευρώπη αποτέλεσε λιμένα ανάπτυξης και ασφάλειας και ε, ε, οι σκαπανείς του ευρωπαϊκού προγράμματος ε, θα ήταν ευτυχείς να δουν αυτήν την πρόοδο. Τώρα, 60 χρόνια μετά την ιδρυτική συνέλευση είναι η δικιά μας ευκαιρία να προωθήσουμε τα θέματα της ευρωπαϊκής πολιτικής είναι ο καιρός ε, της συνεργασίας. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ε, θα πρέπει να αποθυσαυρίσουμε τα όσα έγιναν τα τελευταία 50 χρόνια και να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα καινούριο πρόγραμμα ε, ε, είναι γεγονός ότι οι πολίτες έχουν την τάση να λησμονούν τα όσα έχει επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να τους τα θυμίσουμε. Θα πρέπει να δώσουμε μια νέα πνοή και μια νέα ορμή ε, σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανα της ε, ε, να είναι πιο κοντά ε, στον πολίτη, να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους πολίτες να ολοκληρώσουν, να εκπληρώσουν μάλλον τα οράματά τους και τις επιθυμίες τους. Τα τελευταία συμβάντα έχουν χαράξει όλους μας και γι' αυτό ακριβώς ε, λέμε ότι αυτή τη στιγμή ε, περισσότερο από ποτέ η έκκληση να είμαστε κοντά στους πολίτες έχει μεγαλύτερη ε, σημασία η Μάλτα είναι αποφασισμένη να συμβάλλει στο ευρωπαϊκό ε, πρόγραμμα. Ε, ευελπιστούμε ότι στη διάρκεια της ε, Προεδρίας μας, μέσω της εργασίας μας και μέσω της συνεργασίας μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει δυνατότερη. Γνωρίζουμε ότι έξι μήνες είναι μικρό χρονικό διάστημα. Ωστόσο, Είμαστε φιλόδοξοι και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε ε, στοιχεία του ευρωπαϊκού προγράμματος ε, και ε, να κάνουμε πιο πιστευτή όλη αυτή την ευρωπαϊκή διαδικασία. Θα συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με όρους ειλικρίνειας και εντιμότητας. Όλοι οι υπουργοί ε, ακόμα και οι αρχηγοί της αντιπολίτευσής μας ε, είναι ε, μέλη παλαιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επομένως γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη σημασία που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς επίσης και την σημασία που έχετε εσείς ο καθένας ξεχωριστά ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι εκπροσωπείτε τους πολίτες. Είμαστε περήφανοι που αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κυρίαρχη αρχή η οποία θα μας οδηγήσει ε, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει νέα ορμή ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα πρέπει να γίνει αυτή η εργασία, αυτή η προσπάθεια που θα φέρει τους πολίτες πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα φέρει πιο κοντά και όλους τους εμπλεκόμενους η ασφάλεια, η ενιαία αγορά, η μετανάστευση, ε, η πολιτική ε, ε, γειτονία είναι θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, διότι πιστεύουμε ότι οι πολίτες έχουν πραγματική βασικούς προβληματισμούς ε, στους οποίους θα πρέπει ε, να απαντήσουμε. Δεν θα ασχοληθώ με κάθε μία από αυτές τις προτεραιότητες, ε, αλλά ο Πρωθυπουργό στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο θα αναφερθεί ανελτικά σε όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Μωράες, εγώ θα μιλήσω μονάχα για το πρόγραμμα εργασίας για θέματα που αφορούν την δικιά σας Επιτροπή κυρίως ε, τα θέματα ε, ε, εσωτερικής πολιτικής και τα εσωτερικά ζητήματα τα οποία μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην εργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να φέρουμε κοντά ε, ε, και να προσεγγίσουμε τον κοινό στόχο ε, όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολλά διακυβεύματα και προκλήσεις στον τομέα αυτό. Είναι ένας τομέας όπου πρέπει να επαγρυπνούμε κάθε στιγμή, κυρίως όταν αναφερόμαστε σε θέματα μετανάστευσης και στην απειλή της τρομοκρατίας. Όσον αφορά αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα, ε, πραγματικά είναι δύσκολη και προκλητική η καιρή που περνάμε διανύουμε περίοδο γεμάτη προκλήσεις ε, και για τα κράτη-μέλη και για τα θεσμικά όργανα. Για να μπορέσουμε να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα προς την σωστή κατεύθυνση θα πρέπει να συνεργαστούμε. Ε, ε, η πρόκληση, το διακύβευμα της μετανάστευσης και η απειλή της τρομοκρατίας θα βρίσκονται στο προσκήνιο στη διάρκεια του εξαμήνου. Βασιζόμενοι βεβαίως σε την πρόοδο η οποία έχει γίνει καθώς επίσης και την εμπειρία μας του 2016, κατά τη διάρκεια του οποίου μεγάλα κύματα μεταναστών αντιμετωπίσαμε. Χρειάζεται βεβαίως να αναλυφθούν ε, δράσεις, ε, μακροπρόθεσμες μάλιστα. Η μετανάστευση θα αποτελέσει επομένως μία από τις κύριες προτεραιότητες της Προεδρίας της Μάλτας και θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο ε, ζητήματα που άπτονται του μεταναστευτικού. Θέλουμε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση. Οι 7 προτάσεις οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι και οι οποίες θα οδηγήσουν σε ε, μεταρρύθμιση του κοινού συστήματος ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν σημαντικό τμήμα της εργασίας μας. Εργασίας που έχει ξεκινήσει ήδη και που θα, θα προσπαθήσουμε μέσω των συγκεκριμένων προτάσεων να προωθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Όσον αφορά την προτινόμενη ε, υπηρεσία για το άσυλο, την ΕΑΣΟ, να σας πω ότι έχουμε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να συνεργαστούμε και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε ε, η νέα υπηρεσία να είναι αποτελεσματική και να είναι σε θέση να παράσχει την απαραίτητη αρρωγή. Ε, η πρόταση της Eurodac θα προχωρήσει στο Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο. η Μαλτέζικη Προεδρία θα προσπαθήσει ε, να προωθήσει όσο γίνεται περισσότερους φακέλους ε, που άπτονται του συστήματος ε, ασύλου. και ευελπιστούμε να τα προωθήσουμε αποτελεσματικά. Δυνατότητες για αποτελεσματικά βήματα σε αυτήν την ε, περιοχή, σε αυτό το θέμα, ε, παραμένουν βεβαίως διστακτικά μέχρι ότου καταφέρουμε ε, να απαντήσουμε σε ζητήματα τα οποία αναφέρονται στην συνευθύνη και στην αλληλεγγύη θα πρέπει να προχωρήσουμε λαμβάνοντας υπόψη όσο περισσότερο γίνεται τους προβληματισμούς που έχουν εκφραστεί από διάφορα μέρη. Το θέμα των ετούντων άσυλο ε, ε, δημιουργεί πρόβλημα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως ακόμα περισσότερο την προβληματίζει από ότι τα οικονομικά ζητήματα. Θα πρέπει να μάθουμε από τις διδαχές του παρελθόντος και από τα προβλήματα του παρελθόντος και να διασφαλίσουμε την ύπαρξη των απαραίτητων εργαλείων έτσι ώστε ε, να μπορέσουμε να δουλέψουμε όχι μόνο όταν τα πράγματα είναι εύκολα, αλλά και δυσκολεύουν. Το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου γνωρίζετε ότι συζήτησε ε, το θέμα της ε, δυνατότητας εφαρμογής και του πώς θα εφαρμοστεί η, η αρρωγή και η συνευθύνη και η αλληλεγγύη στο μέλλον. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε συνένεση όσον αφορά την ε, πολιτική ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να τα καταφέρουμε. Έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε ως μέλη ε, μιας ένωσης να ε, επικουρούμε τα άλλα μέλη της ιδίας ενώσεως. Αυτό βεβαίως θα πρέπει να γίνει και μέσω δεσμευτικών αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί από όλους μας από κοινού και βεβαίως θα πρέπει να στείλουμε και το σωστό μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως Προεδρία θα συνεχίσουμε την προσπάθεια υλοποίησης ε, των μέτρων που ε, συμφωνήσαμε ε, ήδη την προηγούμενη χρονιά, έτσι ώστε να βοηθήσουμε ιδιαίτερα στην Ιταλία και την Ελλάδα. Επομένως, ε, θα συνεχίσουμε την εφαρμογή των αποφάσεων ε, για τα hot spots, ε, για την χρήση εμπειρογνωμόνων, καθώς επίσης και για την επαναπρόθεση. Ε, θα πρέπει να δούμε το ε, ε, θέμα της μετανάστευσης με ολοκληρωμένο τρόπο, αντιμετωπίζοντας βεβαίως και τις εξωτερικές διαστάσεις της μετανάστευσης και του ασύλου. Υπάρχει διαρκής ανάγκη συνεχούς προσπάθειας και συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης της μετανάστευσης. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι όσοι δεν έχουν την άδεια να εισέλθουν ή να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι επιστρέφουν στις ε, χώρες τους. Ε, στα πλαίσια λοιπόν αυτά θα πρέπει να ενεργοποιηθούν σωστά οι διαδικασίες ε, της επανεισδοχής και της απομάκρυνσης. Όσον αφορά τις τρίτες χώρες, ε, θα συνεχίσουμε ε, την εργασία όσον αφορά την ε, οδηγία για την μπλε κάρτα για τους πολίτες τρίτων χωρών και θα συνεχίσουμε επίσης και την πολιτική μας για, την, για τις θεωρήσεις βίζα θα συνεχίσουμε την συνεργασία με τις ε, τρίτες ε, χώρες. Έχουν, έχει γίνει ήδη πάρα πολύ, ε, έχει γίνει πολύ καλή δουλειά όσον αφορά την, το Migration Compact με τις πέντε χώρες οι οποίες αποτελούν την ύψιστη προτεραιότητα. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τη Λιβύη και άλλες χώρες της Βόρειας Αφρικής γιατί αυτή η συνεργασία είναι απαραίτητη. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην εξωτερική διάσταση της της ε, ε, μετανάστευσης. Ε, γι' αυτό λοιπόν η Προεδρία θα προωθήσει την διάσκεψη της Βαλέτα του 2015 προετοιμάζοντας μια νέα διάσκεψη το 2017. Η διάσκεψη της Βαλέτα αποτέλεσε ένα εξαιρετικό παράδειγμα αγαστής συνεργασίας και επομένως θα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την οδό για να έχουμε αμοιβαία καλά αποτελέσματα γνωρίζουμε ότι έχουν μειωθεί οι ροές, ε, οι μεταναστευτικές, έστω και αν δεν έχουν σταματήσει. Θα πρέπει ε, να ε, συνεχίσουμε έτσι ώστε η συμφωνία όσον αφορά τους διαδρόμους της μετανάστευσης να συνεχίσει καταβάλλονται προσπάθειες για την εξωτερική διαχείριση των συνόρων ε, η σημασία της οποίας έχει καταδειχθεί λόγω και των τελευταίων προσφάτων προβλημάτων ασφαλείας. Βεβαίως ε, θα πρέπει ε, να βρούμε την χρυσή τομή ανάμεσα στους ελέγχους των εξωτερικών συνόρων και την ομαλή ροή στα σύνορα. Ε, θα καταβληθούν προσπάθειες ε, όσον αφορά ε, το σύστημα εισόδου-εξόδου στα πλαίσια του συστήματος ευφυών συνόρων. και θα καλέσουμε τους ε, να συμφωνήσουν για το σύστημα εισόδου-εξόδου μέχρι τον Ιούνιο του 2017 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί ε, για συμφωνία σχετικά ε, με το σύστημα ETIAS ε, για τις πληροφορίες επί των επιβατών ταξιδιωτών. Η Μαλτέζικη Προεδρία θέλει επίσης να κλείσει την ε, ε, τις ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν στο σύστημα ελέγχου ε, μέσω του αιτίας έτσι ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια. Η Μαλτέζικη Προεδρία θα ήθελε να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των μερών μέχρι τον Ιούνιο του 2017 και ευελπιστεί ότι στο δεύτερο μισό του 2017 θα μπορέσουν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η νέα πρόταση για το σύστημα ΣΥΣ θα λάβει προτεραιότητα προκειμένου να αξιοποιηθεί καλύτερα το σύστημα αυτό για την αντιμετώπιση τη απειλή τη τρομοκρατία. Γιατί υπάρχει η απειλή τη θερμοκρατία και έτσι και η απειλή προ την ασφάλεια των πολιτών μα. Βλέπουμε ότι είναι μια πραγματικότητα, το βλέπουμε και τον τελευταίο χρόνο ιδιαίτερω. και αυτό ο φάκελο παραμένει πολύ ψηλά στι προτεραιότητέ μα. Αναγνωρίζουμε ότι το προφίλ τη δημοκρατίας έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον αντιμετωπίζει πολυάριθμες ε, και πολύπλευρες νέες προκλήσεις που απαιτούν και κατάλληλες, ε, ε, κατάλληλα προσαρμοσμένες απαντήσεις. Γι' αυτό θέλουμε και την προσαρμογή της ανανεωμένης αυτής εσωτερικής στρατηγικής και του δικού χωάρτη για την βελτίωση της ανταλλαγής και διαχείρισης πληροφοριών. Παράλληλα, προσβλέπουμε στα αποτελέσματα της ομάδα, ε, ομάδας, ε, της ομάδας μάλλον υψηλού επίπεδου ε, για το ζήτημα αυτό και θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας εντός του Συμβουλίου για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας και για να καταστήσουμε την Ευρώπη πιο ασφαλή. Τέλος, έχουμε την πρόθεση να συνεχίσουμε την συζήτηση για το θέμα του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και φτάνουμε έτσι στο τέλος του κύκλου πολιτικής για αυτό το θέμα που ηγείται του θεματολογίου για την ε, καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος τα τελευταία τέσσερα χρόνια και μετά θα εντάξουμε και συγκεκριμένες ε, προτεραιότητε για τον νέο κύκλο πολιτική στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Θα είμαστε σε θέση να σημειώσουμε πρόοδο σε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα, μόνο να έχουμε και τη στήριξη των κρατών μελών και εάν υπάρχει και καλή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων μα. Προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σα, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδο σε όλε τι πτυχέ αυτέ προ ε, όφελο και προ το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μπέλα. Κύριε Μπονίτσε, σας παρακαλώ μην υπερβείτε το δεκάλεπτο, διότι έχουμε πάρα πολλές και λεπτομερείς ερωτήσεις από πάρα πολλά μέλη της Επιτροπής μας που θα καλύψουν όλους τους τομείς. Κύριε Μωράης, σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω. Να μην υπερβώ το χρόνο που μου αναλογεί. Για μας είναι μεγάλη τιμή που είμαστε ενώπιν της Επιτροπής σας. Έχουμε ήδη προετοιμάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό την Προεδρία μας. Είναι μεγάλη τιμή που τελικά ερχόμαστε στο Κοινοβούλιο. Ξέρετε, δεν το λέω επειδή περιμένετε να το πω. Πραγματικά. Είμαστε πεπισμένοι πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μάλλον θα πρέπει όλοι να λογοδοτούμε. Πολλές φορές γίνεται αντιλήπτο ως τεχνικό το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ε, θεωρούν οι πολίτες ότι τους αφορά άμεσα. Όμως, νομίζω είναι δικό μας καθήκον Ναι. εξηγήσουμε στους πολίτες ότι το πρωταρχικό μας καθήκον είναι να τους βοηθούμε, να διευκολύνουμε τη ζωή τους. για τις εσωτερικές υποθέσεις, για τα θέματα δικαιοσύνης. Συνεχίζουμε το έργο μας, ούτω ώστε να βελτιώσουμε τη ζωή των οικογενειών και των επιχειρήσεων. Είμαι δικηγόρος και με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα ούτως ή άλλως αυτά τα ζητήματα, αλλά όχι μόνο γι' αυτό άπτονται των ε, θεμελιωδών αρχών μιας δημοκρατικής ε, κοινωνίας. Ε, σεβασμός, αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημοκρατία, ισονομία, κράτος δικαίου, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως λέει και η συνθήκη, αυτές είναι οι κοινέ αξίες όλων των κρατών μελών σε μια ε, πλουραλιστική κοινωνία όπου επικρατούν οι αρχές της ισότητας, της αλληλεγγύης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θα πρέπει όλα αυτά να τα θεωρούμε δεδομένα. Πρώτη φορά να λαμβάνουμε την Προεδρία. Προσπαθούμε να εμβαθύνουμε την συνεργασία μας, οικοδομώντας έτσι μια ισχυρότερη Ευρώπη, σεβόμενη τις ιδιαιτερότητές μας είναι πρόκληση και ταυτόχρονα μεγάλη ευκαιρία για μας. τώρα που λαμβάνουμε την Προεδρία. Ιστορικά λειτουργούσε πάντα ως γέφυρα ανάμεσα σε υπήρους και χώρες η Μάλτα. Φέρνοντας εγκύτερα διαφορετικά συστήματα, διαφορετικές παραδόσεις. Αυτό ε, το μαρτυρεί και η γλώσσα μας. Είναι ένας συνδυασμός πολλών γλωσσών. Προβλέπουμε με ανυπομονησία λοιπόν σε στενή συνεργασία και σε ε, επικοδομητικέ διαπραγματεύσει ανάμεσα στα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα θα εστιάσουμε την προσοχή μα σε διάφορα βασικά ζητήματα που θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα. Η βασική προτεραιότητά μας είναι απλή να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή πρόοδο. Αυτό σημαίνει ότι μας περιμένει πολλή δουλειά. Θέλουμε επίσης ο πολίτης να είναι στο κέντρο του θεματολογίου μας ε, για ολόκληρη την Προεδρία. Αρχίζοντας ε, με το Ευρωπαϊκό ε, Γραφείο Εισαγγελίες, προχωρώντας μετά με την οδηγία που μόλις ε, για την οποία μόλις καταλήξαμε σε συμφωνία. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ζητήματα που είναι μεν τεχνικά, αλλά έχουν ιδιαίτερο ειδικό βάρος για τους πολίτες, για την καθημερινή τους ζωή. Και γι' αυτό θα εργαστούμε σκληρά, για να σημειωθεί πρόοδος σε αυτά τα ζητήματα. Πολλά κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει για το σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με εξαίρεση κάποιες λεπτομέρειες που μάλλον θα διευθετηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Κάποια κράτη-μέλη παρόλα αυτά δήλωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν. Θα εγκριθεί με ομοφωνία ο κανονισμός και με σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Μόλις διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει ομοφωνία για το σχέδιο, Προβλέπει η συνθήκη ότι τουλάχιστον 9 κράτη-μέλη μπορούν να αναπέμψουν το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο. Αν ούτε εκεί προ... Ε, προκύψει συμφωνία, τότε δυνάμει του άρθρου 6 της Συνδίκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να εκκινηθεί η διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας. Δεν ξέρω αν είναι μόνο εννέα κράτη-μέλη που θα ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία. Συνεχίζονται οι συζητήσεις και είναι πολύ πιθανό ότι θα συμβεί. Θα είμαστε σε στενή επαφή με το Κοινοβούλιο σε κάθε περίπτωση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας στο Συμβούλιο. Επίσης, προτιμούμε να διοργανώσουμε σε εθνικό επίπεδο μια διάσκεψη για αυτό το θέμα, διότι ε, ένα κρατέο σύστημα Ευρωπαϊκής εισαγγελία είναι κάτι που επιδιώκουμε να έχει ήδη θεσπιστεί μέχρι το πέρα τη Προεδρίας. Για το σχέδιο κανονισμού Eurojust ολοκληρώνει το Συμβούλιο τη Συζητήσεις για το σχέδιο κανονισμού. Δεν έχει σχέση αυτό με το ΕΠΟ. Ε, αυτό έγινε ε, το Μάρτιο 2015, ξεκίνησε το Μάρτιο του 2015 με τη Λετωνική Προεδρία και τώρα το Συμβούλιο προτίθεται να συζητήσει και να διαπραγματευτεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα τη Eurojust. Κατά πολέμηση τρομοκρατία, μέγιστο μέλημα, ύψιστη προτεραιότητα για μα. συμφωνήσαμε για την οδηγία για την καταπολέμηση τρομοκρατία και θα φροντίσουμε να εγκριθεί. Βάσει και το σχεδίο δράση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση τη καταπολέμηση χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων, θα ενισχύσουμε τις συζητήσεις, περαιτέρω συζητήσεις για την εναρμόνιση των διατάξεων για τις κυρώσεις και για τη δίωξη ποινικών αδειγμάτων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση των κρατικών οργανώσεων, επίσης αμοιβή αναγνώριση για τις αποφάσεις για το πάγωμα και την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων. Έπεται και νέα πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το άκρης ε, το σύστημα πληροφοριών δηλαδή για τα ποινικά μητρώα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κάτι που αναμένουμε ότι θα προχωρήσει επικοδομητικά. Επίσης θα παρακολουθήσουμε τα όσα συμβαίνουν με τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία ε, απελευθέρωση των θεωρήσεων. Τα είπατε και σήμερα το πρωί. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που καταλήξατε σε συμφωνία για την αναθεώρηση του τρέχοντος μηχανισμού αναστολής ε, ισχύως ε, και ήταν προϋπόθεση ε, η συμφωνία για να προβούμε σε περαιτέρω απελευθέρωση. Υπερπηδήσαμε το πρώτο εμπόδιο επίσης. Χαιρόμαστε που καταλήξατε σε συμφωνία για την απελευθέρωση για τη Γεωργία. Στην προηγούμενη Προεδρία θέλουμε να το ίδιο να συμβεί και για την Ουκρανία σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ταυτόχρονα θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και στο Κωσυφοπέδιο και στην Τουρκία στο δρόμο που ακολουθούν προς την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Για το διάλογο, ξέρω πώς σας ενδιαφέρει αυτό το ζήτημα. Η Σλοβαϊκή Προεδρία έκανε αξιολόγηση της, ε, των πεπραγμένων ε, για το διάλογο με το Συμβούλιο μέχρι τον Νοέμβριο του 2015 και πέρυσι υποστηρίξαμε την έκβαση του διαλόγου, δηλαδή την ανάγκη που υπάρχει να συνεχιστεί και να αναβαθμιστεί ο διάλογο στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο έχει συμφωνήσει ότι πρέπει να προετοιμάζουμε πολύ καλά το διάλογο και άρα αυτό φροντίζουμε τώρα να προετοιμάζουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται το διάλογο για να είναι και χρήσιμος. Είναι σημαντικό να είναι κοινό ο στόχο του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Έτσι δείχνουμε έμπρακτα τη δέσμευσή μα για την ενίσχυση του κράτου δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Ελπίζω να έχουμε την αμέριστη υποστήριξή σα. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν διχογνωμίε, Όμω αν συνεργαστούμε μπορούμε να επιτύχουμε σημαντική πρόοδο για του πολίτε, για τι επιχειρήσει, για την κοινωνία μα. Πρέπει να δείξουμε στην Ευρώπη ότι ο στόχος μας είναι να κάνουμε κάτι που θα κάνουμε πραγματικά διαφορά στην καθημερινή του ζωή. Δράτω την ευκαιρία για να επισημάνω ότι είμαστε αποφασισμένοι να, ε, να λάβουμε αυτό το διαμεσολαβητικό ρόλο με πάσα ειλικρίνεια, όπως και στο παρελθόν, για να εκπληρωθούν οι προτεραιότητες στρατηγικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε στενότατα με το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπονίτσι. Ξέρω πόσο έχετε ήδη εργαστεί προετοιμάζοντας ε, την Προεδρία σας. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και εσάς και το επιτελείο σας. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τις ε, ερωταπαντήσεις. Έχουμε και μια έκτακτη ε, συνεδρίαση των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Επομένω, ε, ε, θα δώσω την Προεδρία σε συνάδελφο. Στην κυρία Γκάλ. Έχουμε καταγράψει τη, όσο έχουν στο λόγο ε, και στη... θα αναλάβει λοιπόν η κυρία Γκάλ την Προεδρία από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργή, σα ευχαριστώ για την παρουσίαση σα σήμερα. Η Μορτέζικη Προεδρία είναι μια πολύ περήφανη στιγμή για τη χώρα μου και ε, δικαιώνει και όλου ε, του πολίτε ε, που πίστευαν πριν από τόσα χρόνια ότι θα μπορούσαμε με επιτυχία να συμμετάσχουμε στην Ευρώπη παρά τη γεωγραφική μας θέση και τις αντιδράσεις για την εποχή. Προς τον κύριο Ραβέλα έχω ε, τη, ε, ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση και τη σχετική αναθεώρηση. Είστε ικανοποιημένο. Ε, θέλετε κι εσείς να πιέσουμε για μια Ευρώπη της αλληλεγγύης και της ασφάλειας, όπως είπατε, όπου η ευθύνη είναι επιμερισμένη μεταξύ των κρατών μελών ποιοι ε, συγκεκριμένοι κανόνε προβλέπονται σε ό,τι αφορά του ασυνόδευτου ανελίκου. Και δεύτερον, προ τον κύριο Μπονίτσι, κύριε Υπουργέ, ποια είναι η πρόθεσή σα σε ό,τι αφορά τον ε, φάκελο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το αναφέρατε, αλλά πιο συγκεκριμένα, πού θέλετε να κινηθεί αυτό ο φάκελο κατά τη διάρκεια τη Προεδρία σα. Και επίση, για να είμαι ειλικρινή, σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο για τα έγγραφα του Παναμά. Ένα από τα βασικά προβλήματα ε, του κόσμου στη Μάλτα είναι η διαφθορά. Και όχι μόνο στη Μάλτα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ποιες προτάσεις εσείς θα υποβάλλετε λοιπόν ε, ως Μαλτέζικη Προεδρία για να διασκεδάσετε τις ανησυχίες ε, του Μαλτέζικου λαού αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών αν Ευχαριστώ κυρία Σίπελ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να προσθέσω κάτι στο ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής σε ό,τι αφορά την ευθύνη και την ε, αλληλεγγύη. Γιατί εδώ υπάρχει ε, σημαντικό χάσμα μεταξύ των κρατών Και θα ήθελα η Μαλτιστική Προεδρία να μου εξηγήσει πώς ακριβώς ε, θα προχωρήσει, ούτως ώστε να συμμετάχουν στη διαδικασία περισσότερα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι είναι μάλλον κοινικό που κάποια κράτη-μέλη δεν διαφωνούν ενδεχομένως ανοιχτά ε, στην ε, υποδοχή προσφύγων, όμως ουσιαστικά ε, δημιουργούν τέτοιες τόσο απαράδεκτες συνθήκες που δίνουν και έναυσμα στους πρόσφυγες να φύγουν από τη χώρα αυτή. Εάν δεν τους δίνουμε λοιπόν τη δυνατότητα να ζήσουν αξιοπρεπώς, να εργαστούν, σαφώς και θα φύγουν από αυτή τη χώρα. Ταυτόχρονα όμως μιλούμε για ένα νέο σύστημα ασύλου ε, που προβλέπονται κυρώσει κατά προσφύγων που δεν μένουν στη χώρα στην οποία θα έπρεπε να μείνουν. Πρέπει να το εξετάσουμε λοιπόν αυτό. Ταυτόχρονα έχουμε μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση και εξαιρετικά λυπηρή. Βλέπουμε ανθρώπους να πεθαίνουν στην Ευρώπη, να πεθαίνουν από το κρύο, να ζουν ε, σε σκηνές χωρίς καμία θέρμανση. Και δεν μιλούμε για κάποιες τριτοκοσμικές χώρες κάπου στον κόσμο, μιλούμε για χώρες ε, της Ευρώπης και γνωρίζουμε ε, ότι διαφέρει η οικονομική κατάσταση σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως είναι πια τόσο αδύνατον να συμφωνήσουμε τουλάχιστον να τους δώσουμε κάποια ε, αξιοπρέπεια, να τους παρέχουμε τα ελάχιστα λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται στην Ευρώπη. Ε, ποια είναι η πολιτική σας λοιπόν στρατηγική ε, για να συμμετεχουν προσθετερα περισσότερα κράτη-μέλη στο σεβασμό κάποιων θεμελιωδών, στοιχειωδών ε, αρχών ανθρωπιστικών ε, προτύπων. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τρίτες χώρες, συμφωνώ απολύτως ότι είναι κάτι το απαραίτητο. Θα ήθελα να μου πείτε περισσότερο, περισσότερα για τα κριτήρια ε, συμφωνίας συνεργασίας με τρίτες χώρες και τι είδους συνεργασία θα θέλατε εσείς να δείτε και πώς μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη αποδοχή από χώρες ε, προέλευσης ε, για να ε, υποδεχθούν εκ νέου τους πολίτες τους που δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρώπη. Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συμπληρώνοντας την ερώτηση της κυρίας Μέτσολα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα θέλαμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ στο Κοινοβούλιο. Όμω, βέβαια, δεν έχει κανένα νόημα να δημιουργήσουμε έναν νέο οργανισμό εάν ε, δεν προσφέρει κάτι επιπλέον. Εσείς ε, είστε αισιόδοξοι ότι τελικά θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα με τα κρατημέλη που θα έχει προσταθεμένη αξία. Επιπρόσθετα των όσων ε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ε, κυρίους υπουργούς που ήρθαν σήμερα εδώ ε, να μας ε, μιλήσουν. Σας ευχαριστώ και για όλη αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων που είχαμε μέχρι τώρα, αλλά και που θα έχουμε από εδώ και στο εξή. Συγχαίρω και τη Μάλτα που ανέλαβε την Προεδρία σε μια δύσκολη και αποφασιστική στιγμή για την Ευρώπη. Τώρα βασιζόμαστε σε εσά και βλέπουμε ε, την Μαλτέζικη Προεδρία ως ε, μια νέα ευκαιρία σε ό,τι αφορά την αλλαγή και τον εξυγχρονισμό του κοινού ευρωπαϊκού ε, συστήματος ασύλου, που είναι κάτι που το χρειαζόμαστε τόσο πολύ και οι πολίτες περιμένουν από την Ευρώπη αυτά αποτελέσματα. Επομένω, εκτιμούμε την ε, προσπάθεια που έχετε καταβάλει και την αποφασιστικότητα την οποία έχετε εκφράσει. Τώρα, αναφέρθηκαν συνάδελφοι στο προσφυγικό. Θα ήθελα ε, να πω κάτι ε, ακριβώς όπως είπε και η συνάδελφος προηγουμένως, πώς θα τους δώσουμε πραγματικές ε, ευκαιρίες αυτούς τους ανθρώπους να ζήσουν αυτόνομα και με αξιοπρέπεια για να μην έχουμε και τις ε, δευτερογενείς μετακινήσει στη συνέχεια που είναι ένα από τα βασικά ζητήματα στην πρόταση. Όμως υπάρχουν και άλλα θέματα. Το σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών Schengen. Θα ήθελα να είμαι πολύ ειλικρινή. Η ζώνη Σέγγεν είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα και ήδη εδώ και πολλά χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μας απασχολεί ιδιαίτερως το καθεστώς ε, της Μάλτας ε, ε, για τη χορήγηση διαβατηρίων με καταβολή χρηματικού ποσού. Και βάσει ενός άρθρου πάνω από 700 άτομα έχουν λάβει ευρωπαϊκή ηθαγένεια μέσω της Μάλτας με αντάλλαγμα επενδύσεις και δωρεές στη Μάλτα. Και οι περισσότερες αφορούν πολίτες ε, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της ε, Μέσης Ανατολής. Υπάρχει και ένα άλλο καθεστώς τώρα που αφορά τους Κινέζους ε, πολίτες, που και πάλι αφορά επενδύσεις στη Μάλτα. Όταν θέλουμε να θίξουμε το θέμα και να αντιμετωπίσουμε το θέμα της μετανάστευσης και του προσφυγικού, και αντιμετωπίζουμε τέτοια δυσκολία στο να προσφέρουμε εξωπρεπεί συνθήκε διαβίωση σε αυτού του ανθρώπου, ε, μα φαίνεται μάλλον ηρωνικό να υπάρχει αυτό το φαινόμενο ακόμα στη Μάλτα. Και δεν θέλω να σα κατακρίνω. Θα ήθελα όμω να μα πείτε πώ είναι δυνατόν να συνεχίζετε με αυτή την πολιτική όταν βλέπουμε την ανάγκη ε, για συγκεκριμένου ανθρώπους να φτάσουν με ασφάλεια στην Ευρώπη για να σωθούν και για να έχουν μια νέα ευκαιρία στη ζωή. Ίσως δεν είναι η σωστή προτεραιότητα να δίνεται λοιπόν αυτή η επιλογή ε, σε ε, υπηκόους της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και σε εξαιρετικά πλούσιους Κινέζους πολίτες. Επιστρέφω λοιπόν στην αποφασιστικότητά σας και στις προτεραιότητές σας. θέλω λοιπόν να συνεργαστούμε στενά για το κοινό σύστημα σύλλου και για το Δουβλίνο. Ε, πραγματικά θα ήθελα και εγώ να σας βοηθήσω όσο μπορώ ε, και για το σύστημα ΣΥΣ. Αλλά και για επίσημες και ανεπίσημες ανταλλαγές απόψεων επ' αυτού. vielen Ευχαριστώ. Θα ήθελα κι εγώ να σε ευχηθώ καλή επιτυχία για την Προεδρία σας και θα ήθελα να είμαι ειλικρινής. Ε, έχουμε πολλές ελπίδες, πολλές προσδοκίες να συνεχίσετε και ενδεχομένως να ολοκληρώσετε και κάποια ζητήματα. Ε, φυσικά θα σας υποστηρίξουμε αν δράσετε και εσείς αποτελεσματικά. Ερωτήσεις. Φυσικά σε σχέση με την ε, πολιτική ασύλου και μεταναστευτική πολιτική, ε, είπατε ότι θέλετε να είναι αλληλέγγυα η πολιτική, να υπάρχουν καλύτερες σχέσεις με τα κράτη-μέλη. Πολλά υπόθηκαν ήδη για τους πρόσφυγες. Θέλω να μου πείτε τι γίνεται με το Δουβλίνο. Τι, ποια είναι η επιχειρηματολογία τώρα στο Συμβούλιο. Ε, κάντε μια έκθεση πεπραγμένων να υπάρχει η πρόταση από πλευράς τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ε, ορισμένες φορές υπάρχει ανισορροπία και αυτό είναι εφημισμός, ε, μπορώ να πω και παραλογισμός σε σχέση με τις προτάσεις ε, του Συμβουλίου ε, και πώς εφαρμόζεται. Τέλος πάντων, πώς είναι η κατάσταση και εσείς τι κάνετε με τα κράτη-μέλη. Κανένας δεν θέλει να τους ε, υποδεχτεί τους πρόσφυγες. Ε, Επίση, ε, είπατε θέλετε να βοηθήσετε την Ιταλία και την Ελλάδα. Συμφωνούμε κι εμείς με την προσέγγιση. Θέλουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη μεταναστευτική πολιτική πολιτική ασύλου αυτών των δύο χωρών. Αλλά στην πράξη, τι εννοείται. Ξέρετε ότι δεν λειτουργεί παρά μόνο σε πολύ μικρό βαθμό η συμφωνία με την Τουρκία ε, και αυτή η συμφωνία δεν είναι αποτελεσματική όπως τώρα εφαρμόζεται. Οπότε τι σκοπεύετε να κάνετε και... Η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες για την υποδοχή για τη στέγαση των προσφύγων, κυρίως στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Άκουσα σήμερα, θα ε, επιστραφούν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Ε, τώρα αυτό δρομολογείται επιστροφή προσφύγων βάσει του Δουβλίνου. Εσείς ε, θα το επιτρέψετε αυτό ή θα τηρήσετε επικριτική στάση κατά χωρών όπως η Γερμανία. Μετά, για την ε, πολιτική έχουμε το, ε, τη Σύνοδο της Βαλέτα και τις διάφορες συμφωνίες σύμφωνα με επιμέρους αφρικανικές χώρες. Τι πιστεύετε εσείς, ε, γιατί αυτή είναι η θέση της ομάδας μου, ε, το Σουδάν και άλλε τέτοιε χώρες όπου είναι δικτατορικά καθεστώτα. Μήπω δεν θα έπρεπε να συνάπτουν συμφωνίε επιστροφής με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή, εν πάση περιπτώσει, δεν σας ενδιαφέρει και καρφάκι δεν σας καίγεται αρκεί να πάνε πίσω στην Αφρική. Εγώ θα ήθελα να ξέρουμε ποια καθεστώτα σκοπεύετε να συνεργαστείτε και Τελευταίο σημείο που σχετίζεται όμως αυτή τη φορά με τα μέτρα ασφαλείας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο Επίτροπος Πολάκησε υποσχέθηκε να γίνει αξιολόγηση όλων των μέτρων ασφαλείας που υπάρχουν ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να γίνει λοιπόν η αποτίμησή τους. Αυτό θα συμβεί όσον ούπο μας υποσχέθηκε ο Επίτροπος, οπότε σκοπεύετε και εσείς στο Συμβούλιο να προβείτε σε μια τέτοια αξιολόγηση των επισταμένων μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ποια είναι τα σχέδιά σας για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Αγκάλ, σας παρακαλώ, είναι δίλεπτες οι χρονοθερίδες. Δεν θα έχουν άλλο χρονογόρευσης οι συνάδελφοι. Σαργεντίνη. καλωσορίσατε. Μου δόθη η ευκαιρία, η κυρία Αντέλα, τα τελευταία χρόνια να συζητήσουμε πολλές φορές για αυτά τα ζητήματα. Ήταν πάρα πολύ επικοδομητικές συζητήσεις που είχαμε. Ε, και τώρα μου φαίνεται σαν να ακούω την Σλοβακική Προεδρία. Προτάσεις ε, με κατασταλτικά μέτρα. Το προοδευτικό ε, η προοδευτική πτέρυγα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συγκαταλέγω και εσάς σε αυτή, προσπαθεί να βελτιώσει την κατάσταση. Καλύτερους συνοριακούς εσωτερικούς ελέγχους λέτε εσείς, επιστροφές, αλλά δεν μιλάτε για την αλληλεγγύη καθόλου. Εσείς είσαστε μέσα στη μέση, στη Μεσόγειο, είσαστε δίπλα στην Αφρική. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν μιλάμε για τους παράγοντες πουλ, δηλαδή που ελκύουν τους πρόσφυγες, αλλά πού επιστροφής για να τους ε, παραμένουν εκεί που είναι. Εσείς είσαστε εκεί πέρα και σώζετε τους ανθρώπους και ελέγχετε τα ύδατα, είσαστε στην πρώτη γραμμή. Ποιος είναι ο στόχος των προσφύγων όμως, να φτάσουν ε, στην ενδοχώρα. Μιλάμε για ε, περίκλειστες χώρες. Ε, ε, και δεν έχουν καν θαλάσσια σύνορα. Ε, δεν θέλω να ε, εσείς να προστατεύσετε την κεντροανατολική Ευρώπη, την βορειοδυτική Ευρώπη, γιατί αυ... όλες οι προτάσεις αυτό, ε, ε, σε αυτό αποσκοπούν. Εγώ θα ήθελα από εσά να επηρεάσετε αυτές τις θαλάσσιες οδούς, γιατί οι δικές σας υπερηπολίες στη θάλασσα δυσκολεύουν, αν δεν γίνει κάτι. Είσαστε από ένα μικρό νησί, περιβάλλεστε από θάλασσα, είσαστε δίπλα στην Αφρική. Άλλα περιμένω από εσά. Διαφορετικό αφήγημα που να μιλάει για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Αν εσεί τώρα προωθήσετε τη, τα νομοθετικά σχέδια, τα νομοσχέδια που είναι ε, επιτάπητος αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο, δεν θα βελτιώσει ε, τη θέση και το ρόλο της Μάλτας. Καταλαβαίνετε, αυτά δεν είναι υποδέστερα ζητήματα. Είναι η βασική προσέγγιση που υιοθετούμε για τη μεταναστευτική πολιτική. Και ευτυχώ ε, είδα και την πρόγνωση. Δεν έχετε χιόνι, έχετε 13-14 βαθμούς. Για δείτε όμως στην Ελλάδα. Ε, έχει τόσο πολύ χιόνι και εσείς λέτε πρέπει να προωθήσουμε το φάκελο όπως έχει τώρα. Όχι, γιατί θα συνεχίσουν να πεθαίνουν ε, οι παγόπλητες ε, με πρόσφυγες ε, στην Ελλάδα. Πραγματικά εγώ παίρνω αυτή τη δουλειά στα σοβαρά, πάρα πολύ στα σοβαρά και επώδυνα βλέπω ότι επανέρχεται στα κείμενα της Ολλανδικής Προεδρίας και ασχολείται με τη διαφθορά των πολιτικών. Μα τι εικόνα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτή τη στάση. Ευχαριστούμε κυρία Σαρτζεντίνη. Ακούσαμε όλους τους συντονιστές για να δούμε όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους τώρα. Και μετά θα ακούσουμε τους υπαργούς για να κερδίσουμε χρόνο. Θα διαβάσω τα ονόματα για να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Και θα κλείσει και ο κατάλογος ταυτόχρονα. Mr. Mrs. Mrs. Grappini, Mrs. Schlein, Mr. Zdechovsky, Mrs. Spinelli. And I would like to ask you to keep to a very strict time frame, one, one and a half minutes, because otherwise we won't have time to listen to the answers. Για 1,5 λεπτό, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε χρόνο να ακούσουμε τις απαντήσεις. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε και το λόγο ε, στους υπουργούς. Παρακαλώ, κυρία Χόλμα, η πρώτη. Χίλια ευχαριστώ. Υπουργοί, ε, αντίθετα με αυτά που είπε η συνάδελφος Ατζεντίνη, εγώ έχω διαφορετικές ερωτήσεις και είμαι και απόλυτα πεπισμένη ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε λύσεις με τις αφρικανικές χώρες, όχι ε, για ναι, να επιστρέψουν ναι, οι πρόσφυγες στην Αφρική, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξή. Όταν συνάπτουμε συμφωνίες επιστροφής, έχω την εντύπωση ότι Χρειάζεται συνδυασμός βοήθειας προς τα χωριά, προς τις πόλεις προέλευσης αυτών των προσφύγων, γιατί δεν είναι όλοι από εμπόλεμες ζώνες ε, όπου υπάρχουν σοβαρότητα παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, χρειαζόμαστε πρόγραμμα αρρωγής για την υποστήριξη των επιμέρους περιοχών των αφρικανικών χωρών και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ούτω ώστε να ε, μπορέσουμε να στηρίξουμε τις περιοχές. Ε, ο στόχος δεν είναι μόνο η επιστροφή αυτών των ανθρώπων ε, θα λάβετε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερον, κάτι άλλο που με ενδιαφέρει. Επειδή για την ανταλλαγή δεδομένων υπάρχουν όλο ένα και περισσότερα προβλήματα και με τις νέες δρομοκρατικές πράξεις είδαμε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να λάβουν σοβαρότερε δεσμεύσει, ε, ούτω ώστε να, πρόωρα να ανταλλάσσουν αποτελεσματικά τα δεδομένα για την αποτροπή των τρομοκρατικών πράξεων και επιθέσεων. Ε, έχετε εσεί κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σα για να επιτευχθεί σημαντική πρόοδο. Ευχαριστούμε, Νταλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους κυρίους Υπουργούς. Ε, γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η στιγμή για τη χώρα μας και εγώ είμαι από τη Μάλτα. Είναι μια πολύ μικρή χώρα, αλλά και πάλι παίρνουμε πολύ στα σοβαρά αυτή την Προεδρία. Ε, τώρα, ε, κάποια ερωτήματα που αφορούν τις εργασίες σας. Μιλήσατε για την αλληλεγγύη στη μετανάστευση. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε με περισσότερες λεπτομέρειες ποιες είναι οι προτεραιότητες σας, ιδίως ό,τι αφορά την επανεγκατάσταση των 60.000 προσφύγων από την Ιταλία και την Ελλάδα που θα πρέπει να μετακατασταθούν. Ξέρετε ότι δεν ε, πρόκειται να επιτευχθεί ε, η μετακατάσταση όλων αυτών των ανθρώπων, σε αυτόν τον ε, αριθμό τουλάχιστον. Αυτό θα οδηγήσει σε πολλά προβλήματα και τελικά δεν θα υπάρξει έμπρακτη αλληλεγγύη. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό για την Μάλτα. Θα ήθελα επίσης να μου πείτε με ποιον τρόπο προσπαθεί να επιλύσει το ζήτημα αυτό της μετακατάστασης η Μαλτέζικη Προεδρία και ποιοι στόχοι υπάρχουν για την ε, καλύτερη υλοποίηση του σχεδίου μετακατάστασης όπως αναφέρεται στις προτεραιότητες της Προεδρίας. Και ένα ερώτημα προς τον κύριο Μπονίτσι ε, για τον κανονισμό Βρυξέλλες 2 και πιο συγκεκριμένα για τα δικαιώματα των ε, ανηλίκων και τις περιπτώσεις ε, αντιδικιών ε, σε ό,τι αφορά τη διαφωνία μεταξύ του οικογενειακού δικαίου ε, μεταξύ κρατών μελών. Όταν έχουμε μέλη μιας ίδιας οικογένειας που μένουν σε διαφορετικές χώρες. Η Προεδρία λοιπόν πώς προτίθεται να υλοποιήσει πιο αποτελεσματικά τον κανονισμό Βρυξέλλες 2 και να επιταχύνει την ε, διαδικασία αναδιατύπωσής του. Και τέλος, ποια είναι τα κύρια ζητήματα προς αυτό το θέμα που θέλει να θίξει η Μαλτέζικη Προεδρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους δύο υπουργούς. Προς τον κύριο Ορμπέλα έχω ένα ερώτημα. Όπως ξέρετε, η ασφάλεια παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα για τους Ευρωπαίους. Οι πρόσφατες επιθέσεις ε, στο Βερολίνο ήταν ένα τραγικό ακόμα ε, περιστατικό. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την ε, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών γιατί είναι θεμελιώδης αξίας. Το ΣΥΣ2 διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο προς αυτό. Είναι η μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη βάσει δεδομένων ανταλλαγή πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, μπορεί και πάλι να βελτιωθεί και να δίνει περισσότερα μέσα προ τι αρχέ μα και μεγαλύτερη ασφάλεια προ του πολίτε μα. Στου επόμενου μήνε θα εξετάσουμε τη νέα νομική βάση του ΣΥΣ2. Πρέπει λοιπόν να μεριμνήσουμε ε, για την ενίσχυση της ασφάλειάς του, ε, για να ε, παρέχουμε και προστασία δεδομένων υψηλού επίπεδου και να συμπεριλάβουμε και στοιχεία βιομετρικά, για παράδειγμα. Πρέπει ε, να διασφαλίσουμε ότι θα είναι το καλύτερο δυνατό σύστημα για την αποτροπή μελλοντικών τρομοκρατικών επιθέσεων ε, και για την διασφάλιση της ασφάλειας στην Ευρώπη. Πώς ε, θα επιλύσει το ζήτημα λοιπόν του ΣΥΣ 2 η Προεδρία. Και δεύτερον, θα ξεκινήσουν και νέοι τριμερείς διάλογοι για το ΕΑΣΟ. Εμείς θέλουμε έναν ισχυρό οργανισμό ε, με κυρώσει και επιπτώσεις για όσους δεν συμμορφούνται με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Ποιες είναι οι σκέψεις Προεδρίας. Ελπίζω να μπορούμε να βασιστούμε στην ε, ε, Μαλτέζικη Προεδρία να λύσει αυτό το ζήτημα και μακριά από εθνικούς εγωισμούς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λόπες Αγγιλάρη, σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας αλλά και στο επόμενο εξάμενο σίγουρα θα βρεθεί η βούληση συνεργασίας ε, και από την Επιτροπή μας, την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ε, πολύ σωστά είπατε ότι πρέπει να προωθήσουμε το θέμα της μεταναστευτικής ε, πολιτικής, ε, του προσφυγικού και του συστήματος ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από αυτή την άποψη θεωρώ ότι αυτό που έχετε να προσφέρετε εσείς, ε, η επιπρόσθετη αξία λοιπόν, είναι ότι είστε μια χώρα που για πρώτη φορά αναλαμβάνει την Προεδρία. Μια τόσο σημαντική ευθύνη λοιπόν. Αλλά είστε και μια χώρα ε, που έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, το προσφυγικό. Και πάλι όμως εμένεται σε αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Παρότι είστε σχετικά νέο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχετε σημαντικές ευρωσκεπτικιστικές ε, τάσεις και κινήματα στο πολιτικό σας προσκήνιο. Είστε λοιπόν σε πολύ καλή θέση ε, να λάβετε θέση εντός του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά αυτό το κενό που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίλυση ε, ζητημάτων όπως είναι το μεταναστευτικό και το προσφυγικό και το σύστημα ασύλου. Το έχουμε δει από πλευράς Κοινοβουλίου. Τώρα δίνουμε περιθώριο ευελιξίας σε ό,τι αφορά τη συνομοθέτηση με το Συμβούλιο. Όμως το Συμβούλιο πραγματικά ε, είναι αντίθετο, αντιστέκεται στην υιοθέτηση αποφάσεων αλλά και στην υλοποίηση των αποφάσεων που έχει υιοθετήσει το Συμβούλιο μέχρι τώρα σε ό,τι αφορά τα επιμέρους ε, επεισόδια της ε, προσφυγική κρίσης. Και αυτό αφορά κάτι πολύ συγκεκριμένο που θα ήθελα να αναφέρω. Και σε αυτό σίγουρα θα επανέλθουμε και στο επόμενο εξάμεινο. Ο κώδικας θεωρήσεων μπλοκάρεται από το Συμβούλιο. Αντιστέκεται λοιπόν, θέτει αντιρρήσεις ε, χωρίς κανένα πνεύμα συμβιβασμού για ανθρωπιστικούς λόγους. Έχετε λοιπόν μια ευκαιρία, μόνο όμως να ακολουθήσετε τις αξίες σας, το ευρωπαϊκό σας πνεύμα, όχι μόνο τις ε, υποχρεώσεις σας λοιπόν αλλά τον πρωταγωνιστικό ρόλο που θέλετε να ε, λάβετε για τα ζητήματα μετανάστευσης ε, και ασύλου. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε τη διαφορά και εγώ εκφράζω αυτή την προσδοκία που έχω ότι θα ξεχωρίσετε και ε, θα κάνετε τα δέοντα για να ξεμπλοκάρουν αυτά τα ζητήματα και να συνεχιστεί ο κώδικας θεωρήσεων με μια νέα νομική οδό που πρακτικά θα σημαίνει ότι θα υπάρχει και ένα περιθώριο ευελιξίας για τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους υπουργού για την παρουσία τους εδώ σήμερα. Δύο ερωτήσεις και ένα σχόλιο. Κύριε Αρμπέλα, είπατε κάτι πολύ σημαντικό για τη μετανάστευση. Θέσατε τη μετανάστευση στο επίκεντρο της πολιτικής σας δράσης κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Όμως, ε, Υπάρχουν και δύο ακόμα ζητήματα που πρέπει να εξετάσουμε. Πρώτον, το θέμα τη ε, ένταξη, τη ενσωμάτωση. Είναι πολύ σημαντικό, θα έπρεπε μάλλον είναι πολύ σημαντικό ε, τμήμα του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματο Ασύλου και μεταναστευτική πολιτική. Γνωρίζω βεβαίω ότι η ενσωμάτωση είναι θέμα των κρατών μελών, Όμω και πάλι χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων και θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο ευρωπαϊκό σύστημα ε, κοινωνικής ενσωμάτωσης. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, για την αύξηση της ριζοσπαστικοποίηση σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε συγκεκριμένα σχέδια για ε, να δοθεί ένα τέλος αυτή την ριζοσπαστικοποίηση στους μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς στην Ευρώπη. Και τελευταίο σχόλιο. Εγώ ως εισηγητής ε, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου, ε, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε απολύτως έτοιμοι για τις διαπραγματεύσεις και με τα χαράς ε, θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις υπό τη δική σας Προεδρία. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμε, καλώ ήρθατε κύριε Υπουργή και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για την Προεδρία. Ήδη αναφέρθηκαν τα έγγραφα του Παναμά και δεν είναι μόνο θέμα διαφθορά. Είναι και θέμα αξιοπιστίας μας. Υπήρχε αυτός ο υπουργός που εμπλεκόταν στο σκάνδαλο για τον εγγράφο του Παναμά και δεν υπήρχε καμία κοινοβουλευτική διερεύνηση. Ε, και μάλιστα θα τεθεί και επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Συμβουλίου. Θέτει λοιπόν και ζήτημα αξιοπιστία. Όμως ε, εδώ έχουμε μια τεράστια προσπάθεια κάλυψης ε, οργανωμένου εγκλήματος ακόμα και δρομοκρατίας. Εδώ εξετάζουμε την πρόταση κατά του ξεπλήματος ε, χρήματος και ε, κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας την οδηγία ΠΥΦ. Ελπίζω να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της Μαλτέζικης Προεδρίας, αλλά δεσμεύεστε πραγματικά ότι θα την ολοκληρώσετε, ότι θα θεσπίσετε μαύρο, μαύρη λίστα φορολογικών παραδείσων όπως προτείνει η Κομισιόν. Πρέπει να καταπολεμήσουμε το ξέπνιμα χρήματος λοιπόν, ε, να αντιμετωπίσουμε αυτές, τους αυτούς μηχανισμούς και τις δομές που μου λένε ότι υπάρχουν στις χώρες σας. Και μετά συνδέεται και με το άσυλο και με την ε, αξιοπιστία του συστήματος Σέγγεν, αλλά και την καταπολέμηση του οργανωμένου ε, εγκλήματος και της τρομοκρατίας. αυτό το IIP, το πρόγραμμα των μεμονωμένων επενδυτών ε, και των χρυσών θεωρήσεων. Εντάξει, δεν είστε μόνο εσεί και η χώρα μου, η Πορτογαλία τα έχει. Όμω σα ρωτώ, θα πιέσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει αυτά τα καθεστώτα. Προφανώ και υπάρχουν. Εντάξει, δεν είναι μόνο ανήθικο ότι σκεφτείτε ότι ε, αποτρέπουμε πρόσφυγες που χρειάζονται στήριξη και εμείς τους αποτρέπουμε από το να έρθουν αλλά είναι εξαιρετικά αρνητικό και για την ασφάλειά μας, γιατί αξιοποιούνται αυτοί οι μηχανισμοί από το οργανωμένο έγκλημα. Θα δώσετε λοιπόν τους καταλόγους των ατόμων που έλαβαν τέτοιες χρυσές θεωρήσεις και έλαβαν καθεστώς IPP, όχι σε εμά, γιατί θα πείτε ότι είναι θέμα προστασίας δεδομένων, όπως λένε και οι πορτογαλικές αρχές. Θα τα δώσετε στη Europol για να ελέγξουν και να μας ενημερώσουν ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Σας καλώ λοιπόν να δώσετε τη λίστα για το 2015 και 2016, ούτως ώστε όντως να ελεγχθούν και στα τέλη της Προεδρίας σας θα δούμε αν υπάρχουν προβλήματα σε αυτές τις λίστες ή όχι. Ευχαριστώ κυρία Κιέγκα. E, ε, σας ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα ε, να ευχηθώ τα καλύτερα στην, ε, στην Προεδρία. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και για τα όσα μας είπατε. Κυρίως γιατί εις το παρελθόν είχαμε πολύ καλή συνεργασία και ευελπιστώ λοιπόν ότι και υπό την Προεδρία της Μάλτας θα συνεχίσουμε αυτή την καλή συνεργασία. Σας ευχαριστώ και για την διαθεσιμότητα ε, που δείξατε όταν ε, ήρθαμε σήμερα φέτος το καλοκαίρι με μια αποστολή της ε, ΛΥΜΠΕ και επίσης μετά από πάρα πολλά χρόνια θα έρθει μια αποστολή των χωρών ΑΚΕ Αφρικής Καραϊβικής Ειρηνικού στην Μάλτα. Οι ερωτήσεις μου στρέφονται κυρίως στον Υπουργό κύριο Αμπέλα συνέχεια των εργασιών του Κοινοβουλίου αναφέρεται, γιατί είπατε ότι θέλετε με ολιστικό τρόπο να αντιμετωπίσετε το, το μεταναστευτικό, που δεν είναι έτσι ένα, μια απλή επικεφαλίδα, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ε, εγώ θα ήθελα να ε, ε, και στην Προεδρία σας να, το, να καταδείξετε ότι πραγματικά το εννοείτε αυτό. Επίσης, συμμερίζομαι πλήρως τους προβληματισμούς σας σε σχέση με την έλλειψη αλληλεγγύης, κυρίως γιατί και οι δυο μας προερχόμαστε από παρόμοιες γεωγραφικά χώρες, δηλαδή είμαστε από χώρες του Νότου και επομένως και από τη δική σας πλευρά περιμένω μεγαλύτερη ευαισθησία έτσι ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε το κοινό μας θεματολόγιο. Ερώτηση, έχετε συγκεκριμένες προτάσεις έτσι ώστε να εφαρμόσετε ε, στην πράξη την αρχή της αλληλεγγύης, θα προτείνετε τροποποιήσεις ε, στον κανονισμό του ε, ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά το κριτήριο της χώρας ε, πρώτης ε, υποδοχής και έχετε την πρόθεση να υποβάλλετε εναλλακτικέ προτάσεις όσον αφορά το relocation. Πώς θα πείσετε τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να υλοποιήσουν τις υποχρεώσεις σας. Τέλος, θα βάλετε στις προτεραιότητες σας μια πολιτική ένταξη στο ευρωπαϊκό έδαφος των μεταναστών και των προσφύγων όσον αφορά τα κοινωνικά κοινωνικά θέματα, γιατί αναφερθήκατε στα κοινωνικά ζητήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, κύριοι ε, Υπουργοί, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ για την ε, Μαλτέζικη ε, Προεδρία. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν ήδη οι συνάδελφοι. Το πρόβλημα της μετανάστευσης και όλα τα άλλα ζητήματα που αναφέρθηκαν βεβαίως είναι πολύ επίκαιρα θέματα και τα και προσυπογράφω. Θα ήθελα εγώ να αναφερθώ σε κάτι άλλο. Αναφερθήκατε στο ευρωπαϊκό σχέδιο, την ανάγκη ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να Ε, και την ανάγκη να προωθήσουμε λοιπόν το πρόγραμμα αυτό. Ε, Πολύ λιγότεροι πλέον πιστεύουν στη χώρα μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως δεν άκουσα μεταξύ των προτεραιοτήτων σας να αναφέρετε ακριβώς αυτό το πρόβλημα της διάσπασης της Ευρώπης ε, λόγω Σέγγεν, της Ευρώπης αυτής που είναι πλέον δύο ταχυτήτων. Αναφερθήκατε στο σεβασμό των συνθήκων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχω την αίσθηση ότι οι πολίτες ε, των χωρών όπως η δικιά μου που δεν ε, συμμετέχουν στο χώρο Σέγγεν ε, αντιμετωπίζουν διακριτική μεταχείριση στις μετακινήσεις τους. Η Ρουμανία όμως έχει πολύ καλό μητρό όσον αφορά την τρομοκρατία ας πούμε. Και σήμερα άκουσα ένα νέο που αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο ε, και αφορά έναν επιπλέον φόρο ε, που θα επιβληθεί στους ε, μετανάστες που προέρχονται από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Μα γιατί αυτή η διακριτική μεταχείριση δεν γίνονται σεβαστείς οι συνθήκες ούτε αυτή τη φορά. Thanks. Dear Minister, I welcome you. Ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω, λέει η κυρία Σλάιν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 Ε, σας καλωσορίζω λοιπόν και τους δύο. Ε, πολλά ενδιαφέροντα μας είπατε. Εδώ συζητούμε για μια πρόταση του, ε, ε, της ε, Κομισιόν και το Συμβούλιο δεν, μας είπατε δεν συζητά επί της ουσίας. Θα ξεκινήσετε τη συζήτηση επί τη βάση της πρότασης της Κομισιόν ή θα συνεχίσετε να συζητάτε επί των εγγράφων της Σλοβακικής Προεδρίας για την λεγόμενη λεγόμενη ε, έννοια της αλληλεγγύης που στην ουσία αποτελούν ε, παρεκφυγές έτσι ώστε να μην ασχοληθούμε με το πραγματικό θέμα της αλληλεγγύης ε, που σημαίνει ότι με αξιοπρεπή τρόπο θα υποδεχτούμε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ε, υποδοχής. Αναφερθήκατε επίσης στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί η αλληλεγγύη και η ε, ευθύνη. Επανειλημμένα ε, έχουμε αναφερθεί στο θέμα αυτό εμείς εδώ και ζητήσαμε το θέμα αυτό εδώ, ε, κυρίως όσον αφορά την υπέρβαση των εμποδίων και των κολλημάτων στην ε, είσοδο. Ε, εμείς πιστεύουμε ότι πλέον όπιστο δρομούμε αντί να προχωρούμε. Θα πρέπει οι χώρες να, να τηρήσουν τα υποσχεθέντα και τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει όσον αφορά τη relocation. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρέπει να μας πείτε αν θα τα προωθήσετε. Ευχαριστώ. Vážení eh, Ευχαριστώ για τι για τις παρουσιάσεις σας, ε, κύριε Υπουργή. Εγώ είμαι ε, μεγάλος οπαδός ε, της Μάλτας. Τις διακοπές μου τις περνάω συχνά στη χώρα σας και παρακολουθώ από κοντά τις εξελίξεις. Θέλω να πω ότι από όλα αυτά που έκουσα με και έμαθα, ε, με απογοήτευσε το εξής. Ε, ε, επισκέφθηκα τα κέντρα κράτησης της Μάλτας. Ευχαριστώ που με υποδεχτήκατε και δεν ήμουν μέλος μιας υπές, επίσημης αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ που με αφήσατε να επισκεφθώ αυτά τα κέντρα Επειδή διαβάζω και τις εφημερίδες σας, Βλέπω ότι ανθεί η διαφθορά στη χώρα σας. Ε, είναι θέμα μεγάλο για σας. Και όντως είναι περίπλοκο αυτό το ζήτημα και ποτέ κανείς δεν θα καταφέρει να εκριζώσει την ε, διαφθορά 100%. Όμως βλέπω ότι έχετε ιδιαίτερο πρόβλημα. Καταλαβαίνω ότι λόγω εγκύτητας με τη Σικελία μπορεί να έχει αυτό αρνητικές επιπτώσεις. Α, να πω και κάτι άλλο. Αναφερθήκατε στο φιλόδοξο ε, σχέδιό σας να εγκριθεί η πρόταση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όμως, ε, έχουμε ήδη απευθύνει πολύ επικριτικά σχόλια προς τη σλαβακική Προεδρία για κάποια ζητήματα. Ο Ευρωπαϊκός εισαγγελέα θα έχει τον ίδιο μισθό με έναν Τσέχο εισαγγελέα. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα πέρα από τα μισθολογικά για τα οποία έχουμε ε, ήδη αποστείλει τέτοια επικριτικά σχόλια και θέλουμε να ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις σας. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές, πολλές ανοησίες μέσα στο σχέδιο επίσης για τα όπλα και τα πυρομαχικά, ε, παραδείγματος χάρη καταγραφή των μικρών πυροβόλων όπλων. Πρέπει να τροποποιήσετε αυτό το σχέδιο και θα δημιουργηθεί χάος στην Ευρώπη και θα γυρίσει μπούμερανγκ αυτό. Ευχαριστούμε, Σπινέλη. Καλωσορίζω τους εκπροσώπους της Μαλτέζικης ε, Προεδρίας, ε, στην οποία ε, πραγματικά βασίζομαι, υπολογίζω πολύ. Οι συμφωνίες ε, της ε, Βαλέτα και η συμφωνία με την ε, Λιβύη αναφέρθηκε προηγουμένως. Ποια είναι η απόψή σας όσον αφορά την χθεσινή αποστολή πολεμικών φρεγατών της Ιταλίας στα χωρικά ύδατα της Λιβύης. Πιστεύετε ότι ε, ελοχεύει κίνδυνος ε, σε σχέση με το, ε, με το θέμα της καταπολέμησης των διακινητών στην Λιβύη. Δεν θεωρείτε ότι εδώ μπορεί να, υπάρξουν, να υπάρξει ένα βίωση μνημών απεικιοκρατίας όσον αφορά την διαδικασία της μπλε κάρτας. Ε, μπορείτε να κάνετε κάτι όσον αφορά την πεισματική θέση του Συμβουλίου απέναντι της ε, προτάσεως ε, της Κομισιόν. Δεν θα πρέπει να προσπαθήσετε να διευκολύνετε κάπως διαδικασίες για την μπλε κάρτα. Τρίτον, σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση, συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία και τα όσα συμβαίνουν στην Λέσβο, όπου λείπουν τρόφιμα, ε, δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση κλπ. Ε, δεν θα πρέπει ε, να το ξανασκεφτείτε, το να σταλούν δηλαδή πρόσφυγες από άλλες χώρες βάσει τη συμφωνία του Δουβλίνου ξανά στην χώρα αυτή και βεβαίως ε, δεν θα πρέπει να το δούμε λίγο και ως ε, έγκλημα ε, διότι παραβιάζονται κατάφορα διεθνείς συνθήκες. Θέλω την άποψή σας επ' αυτού. Χιμένες Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας για την παρουσία σας μάλλον και την παρουσίασή σας. Ε, σε αυτό το σενάριο των ε, απειλών των τρομοκρατικών και αν θεωρήσουμε ότι η τρομοκρατία αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διότι παραβιάζει βασικά θεμελιώδη δικαιώματα, το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην ακεραιότητα, το δικαίωμα στην ασφάλεια των ατόμων, το δικαίωμα στην προστασία, γιατί ε, ξέρετε ότι οι τρομοκράτες ε, σκοτώνουν έναν, αλλά τρομοκρατούν και όλους τους υπόλοιπους. Επομένως είμαστε όλοι ε, θύματα, αλλά τα πραγματικά θύματα της τρομοκρατίας είναι οι μεγάλοι λησμονημένοι. Λίγα, λίγο καιρό μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα ούτε ξέρουμε τι κάνουν και όλοι τους ξεχνούν. Ε, εγώ επί χρόνια ζητώ να υπάρξει οδηγία για τα θύματα της τρομοκρατίας, γιατί πιστεύω ότι είναι πράγματι απαραίτητη. Εμείς ε, έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε ε, πολλές προσπάθειες ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε και οδηγία για τα θύματα της τρομοκρατίας και οδηγία για τα θύματα του, του τράφικινγκ ε, και ε, δεν ξέρω ποια είναι ακριβώς το, τα εργαλεία τα πιο ενδεδειγμένα, αν θα πρέπει να είναι οδηγία ή κανονισμός, αλλά θα ήθελα πραγματικά να υπάρξει κάτι ε, και θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό. Πολλές ερωτήσεις, λέει η Προεδρεύουσα, έχετε. Αγαπητοί υπουργοί, μπορώ να σας δώσω από 10 λεπτά στον καθένα για τις απαντήσεις. Ε, γιατί πραγματικά δεν έχω περισσότερο χρόνο. Ήταν πολλέ οι ερωτήσεις. Ε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Αμπέλα προηγουμένως. 10 λεπτά για σας και 10 λεπτά για τον κύριο Μπονίτσι. like to... Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις ερωτήσεις σας. Βεβαίως ε, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και επίκαιρες ερωτήσεις. που απευθύνεται και σε μένα προσωπικά σε ό,τι αφορά το θέμα της μετανάστευσης. Όπως ξέρετε, το θέμα της μετανάστευσης έχει συζητηθεί επί μακρόν. Τουλάχιστον τώρα αναγνωρίζουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει και να επιληθεί από τις ευρωπαϊκές χώρες συνολικά. Όμως αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση, όπως εξήγησα και στην ε, εισήγησή μου. Και η βάση της συζήτησης αυτή σίγουρα είναι η αλληλεγγύη. Γι' αυτό και αναφέρθηκα στην αρχή της αλληλεγγύης ε, προηγουμένως. Και σίγουρα είναι ο κοινό ε, τόπος πάνω στον οποίο θα βασιστεί αυτή η συζήτηση. Επίσης, ανέφερα και σήμερα, αλλά και στο παρελθόν, ότι πρέπει να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση ως προς τη μετανάστευση. Για να επιτύχουμε τη σύσταση ενός ε, κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου δεν είναι ένα μεμονωμένο θέμα που πρέπει ε, να εξετάσουμε. Πρέπει να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση λοιπόν ως προς τη μετανάστευση. Και όπως είπα βέβαια και η ελληνική είναι πολύ σημαντική και η ευθύνη ε, πάει χέρι-χέρι με την ελληνική. Δεν χρειάζεται να δώσουμε ορισμό για την αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι η αλληλεγγύη. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να εξετάζουμε τις συζητήσεις που έχουν λάβει η χώρα και υπό τη Σλοβακική Προεδρία Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορές στο Συμβούλιο και ο ρόλος της Προεδρίας είναι να γεφυρώσει αυτές τις ε, διχογνωμίες, τις διαφορές απόψεων, την προσέγγιση του μεταναστευτικού γι' αυτό πιστεύουμε πραγματικά ότι πρέπει να υπάρξει ολιστική προσέγγιση και να έχουμε κατά νου και την εσωτερική και την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης. Σίγουρα, αυτό που σας απασχόλησε ιδιαίτερος ε, και αναφέρατε και πολλά, πολλές ερωτήσεις προς αυτό, ε, είναι η αναθεώρηση του Δουβλίνου. Αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του Δουβλίνου Επίσης αναγνωρίζουμε ότι οι ισχύοντες ε, κανόνες που έχουν θεσπιστεί εδώ και πολλά χρόνια πλέον ε, δεν είναι κατάλληλοι για την διαχείριση του μεταναστευτικού ε, πλέον, όταν έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες που διέρχονται στην Ευρώπη σήμερα. Η οδός της Κεντρικής Μεσογείου είναι η πιο διαδεδομένη. Αυτό είδαμε πέρσι, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη διέλευση, αλλά δυστυχώ και τον αριθμό των θανάτων. Γιατί βέβαια εδώ δεν μιλούμε για αριθμητικά στοιχεία, για νούμερα, μιλούμε για ανθρώπινες ζωές. Η μετανάστευση έχει και ένα ανθρώπινο πρόσωπο και θα πρέπει πάντα να το θυμόμαστε αυτό. όταν ε, εξετάζουμε τη διαχείριση του προβλήματος ε, και τις λύσεις που θα δώσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σωστά αναφέρατε το θέμα της ε, επανεγκατάστασης και είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει ως κράτη-μέλη. Πρέπει όντως να τηρούμε τις αποφάσεις τις οποίες υιοθετούμε και να τις υλοποιούμε. Αυτό είναι και ένα τεστ αξιοπιστίας και για εμάς τα κράτη-μέλη αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη. Όντως, λοιπόν, θα πρέπει να συνεχίσουμε το διάλογο και να καλούμε τα κράτη-μέλη να τηρούν τις δεσμεύσεις τους. Και αυτό είναι σημαντικό για τη διαχείριση και επίλυση του μεταναστευτικού ζητήματος, ιδίω όταν τα κράτη-μέλη βρίσκονται υποποίηση. Και όπως ε, σωστά αναφέρατε, η Ιταλία και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι οι χώρες οι οποίες ε, ε, αναφέρεται και αναγνωρίζεται ότι χρειάζονται μεγαλύτερη βοήθεια. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ε, για το θέμα της μετανάστευσης και να... θα είναι δύσκολη η επίτευξη συμβιβασμού, δεν είναι εύκολο καθήκον, σίγουρα, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια, τον πολιτικό διάλογο και η βάση του διαλόγου να είναι η ευθύνη και η αλληλεγγύη και ότι είμαστε μαζί σε αυτή τη διαδικασία άμεσα ή έμεσα όλα τα κράτη-μέλη επηρεάζονται από το φαινόμενο της μετανάστευσης. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού. Μετά υπάρχει και το θέμα των τρίτων χωρών και των χωρών διέλευσης. Η σύνοδος της Βαλέτα ήταν πολύ σημαντικό ορόσημο θεωρώ όταν είχαμε τους Αφρικανούς και τους Ευρωπαίους ηγέτες ε, συμφωνήσαμε επί ενός ε, σχεδίου δράσης το οποίο και πάλι θα πρέπει να υλοποιηθεί. Γι' αυτό και εισηγητικά είπα ότι θα έχουμε μία ε, συνεδρίαση ε, υψηλού επίπεδου στις αρχές Φεβρουαρίου για να γίνει μια αποτίμηση της κατάστασης. Σημαντικό είναι να μειώσουμε τον αριθμό των μεταναστών που φεύγουν από τις χώρες τους. Όμως θα πρέπει να βοηθήσουμε και τις τρίτες χώρες να αναπτυχθούν περαιτέρω, ούτως ώστε να μην φεύγουν οι πολίτες τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, παράλληλα, θα πρέπει και να προστατεύουμε, να δίνουμε καταφύγιο σε όσους το δικαιούνται και σε όσους ε, μπορούν ε, να λάβουν το καθεστώς του πρόσφυγα. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει γρήγορα να προχωρούμε στην επανεισδοχή όσων ε, δεν δικαιούνται διεθνούς προστασία, διεθνή προστασία. Είναι σημαντικό λοιπόν να εξετάσουμε την πολιτική κατάσταση και την έλλειψη σταθερότητα στην ε, Βόρεια Αφρική. Αναφέρθηκα ιδιαίτερω ε, στη Λιβύη, αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Όντω, ε, η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία είναι σημαντική και θα πρέπει να γίνεται σεβαστή. Ιδάλω θα έχουμε μεγαλύτερη εισρωή μεταναστών προς την Ευρώπη με όλες τις δυσκολίες που αυτό συνεπάγεται. Όμως θα πρέπει να εργαστούμε από κοινού σε ό,τι αφορά το θέμα της μετανάστευσης. Τώρα, περνώ στο θέμα της ασφάλειας. Σαφώς και υπάρχουν ε, απειλές. Γνωρίζετε κι εσείς ότι η άρση των ε, εσωτερικών συνοριακών ελέγχων απαιτεί ομοφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μέχρι τότε πρόθεση της Προεδρίας είναι να βελτιώσουμε κατά το δυνατόν την πρόσβαση ε, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ε, στα σχετικά συστήματα ε, και στο σύστημα εισόδου του ΣΥΣ. Και η ριζοσπαστικοποίηση ήταν από τα θέματα που αναφέρατε. αξίζει να σημειωθεί ότι ε, υπάρχει και το δίκτυο επίγνωσης της ριζοσπαστικοποίησης που λειτουργεί καλά και θα πρέπει να το ενισχύσουμε. Όμως ε, μας απασχολεί ιδιαίτερα και το θέμα της επιστροφής ε, των νέων. Κάποιοι από αυτούς έχουν γεννηθεί σε περίοδο σύγκρουσης. Μας προβληματίζει αυτό και θα πρέπει λοιπόν να τους επανεντάξουμε και να τους στηρίξουμε. Πέραν τούτου λοιπόν, συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου ε, και των ε, μυστικών υπηρεσιών θα πρέπει να συνεχιστεί. Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών ε, είδαμε μια βελτίωση. Θα πρέπει λοιπόν να βασιστούμε σε αυτό το θετικό βήμα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, αλλά και να ενεργήσουμε περαιτέρω. Ανταλλαγή πληροφοριών λοιπόν, αλλά και ανάληψη δράσης με βάση αυτές τις πληροφορίες. Νομίζω λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας, έχουμε τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων, με το σύστημα ΣΥΣ, όπως αναφέραμε, Είχαμε πρόσφατα και την ε, δημοσίευση της Επιτροπής για το ΣΥΣ2. Θα γίνει και η σχετική συζήτηση. Ουσιαστικά και εμείς θέλουμε περισσότερη ασφάλεια για τους πολίτες μας, περισσότερη ασφάλεια για την Ευρώπη. Είναι, ε, υπάρχει σημαντική ανησυχία για τους πολίτες μας. Και πολύ σωστά αναφέρατε κι εσείς. Όταν βρισκόμαστε κοντά στους πολίτες, όπως ε, βρίσκομαι εγώ, γνωρίζετε ότι η τρομοκρατική απειλή είναι ένα σημαντικό, μια σημαντική πηγή ανησυχία στους πολίτες μας. Θα μας απασχολήσουν πολλά αυτά τα θέματα της ασφάλειας, ε, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της μετανάστευσης βεβαίως. Θα εξετάσουμε μια σειρά προτάσεων, όμως θα πρέπει να ε, είμαστε υπεύθυνοι και αλληλέγγυοι. Αυτή θα είναι η βάση της συζήτησής μας. Ευχαριστούμε κύριε Μέλα για τις απαντήσεις σας. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Μπονίτσι. Thank you very much for your... Ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Πολλές ερωτήσεις σχετίζονται με τις προθέσεις της Προεδρίας και με ρωτήσατε και για κάποια τοπικά χώρια ζητήματα. Ως ε, Προεδρεύον του Συμβουλίου Υπουργών ε, Δικαιοσύνη, θα ήθελα να σα απαντήσω κατά προτεραιότητα για αυτά τα ζητήματα που σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο μου. ΕΠΟ, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι ένα μέσο αποτέλεσμα συμβιβασμού και Κάποιοι ε, συνάδελφοι υπουργοί μου είπαν δεν επαρκεί, ε, δεν επαρκούν διατάξεις για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, άλλοι μου λένε το αντίθετο. τι να πω, είναι συμβιβασμός. Κάποιοι πιστεύουν ότι στερεί, κάποιοι ότι είναι υπερβολικό αυτό το μέσο. Όλοι έχουν τις δικές τους απόψεις, το ίδιο και εγώ. Τώρα όμως, επειδή κρατάει χρόνια η συζήτηση για το ΕΠΟ, τα τρία-τέσσερα χρόνια στο Συμβούλιο, τα τρία-τέσσερα τελευταία χρόνια συζητούμε το θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Συμβούλιο. Και τώρα ε, είναι κάποια κράτη-μέλη που είπαν «Ε, δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε. Ε, λοιπόν, ωραία, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Καταγράφουμε ότι δεν υπάρχει ομοφωνία και ε, θα πρέπει να διαπιστώσουμε στη συνέχεια αν υπάρχουν κράτη-μέλη που θέλουν να προχωρήσουν επί τη βάση μιας ενισχυμένης συνεργασίας. Αν συμβεί αυτό και πιστεύω ότι θα συμβεί, Ο ρόλος της Προεδρίας στη σύνδεση των Υπουργών Δικαιοσύνης είναι να το προωθήσουμε. Και αναλαμβάνω δέσμευση ενώπιόν σας. Ε, θα ε, μεσολαβήσω, θα διευκολύνω αυτή την πρωτοβουλία. Προβλέπετε αυτό στη συνθήκη. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν, οπότε στο μέτρο του δυνατού θα ε, διευκολύνουμε εμείς τη διαδικασία για να συγκροτηθεί το γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη δέσμευση. Άλλη δέσμευση. Συνεργασία στενή με το Κοινοβούλιο. Πρέπει να μας βοηθήσετε. Μαζί θα τα καταφέρουμε αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θέλω το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να συνεργαστούν. Τρομοκρατία. Μετά μου είπατε για την τρομοκρατία. Φυσικά. Είναι στον πυρήνα των ανισχυών που έχουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν με τον κύκλο όμως. Υπάρχουν αυτά τα μέτρα. Επιδιώκουμε την εφαρμογή τους. Κυρίως για τον ε, οδικό χάρτη για την ανταλλαγή και διαλειτουργικότητα που εγκρίθηκε πέρυσι και η οδηγία PNR. Επίσης, πρόληψη και καταπολέμηση της δροσπαστικοποίησης ε, και της βίας ε, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Είμαι επίση υπεύθυνο ε, και για τα πολιτιστικά ζητήματα. Να συζητήσουμε την οδηγία για τα οπτικοακουστικά. Ε, λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της συζήτησης, όταν μιλάμε για ρητορική μίσους ε, και για ριζοσπαστικοποίηση και το ρόλο των ε, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όλα αυτά θα δεληφθούν υπόψη ε, και θα τα συνδυάσουμε με την ε, μεταξέλιξη του συστήματος πληροφοριών του Σέγγεν και με την Συμφωνία Πρώτης Ανάγνωσης για την Οδηγία για την Καταπολέμηση της ε, Τρομοκρατίας. Η Συμφωνία είναι φρέσκια από τον περασμένο μήνα και αν, γίνεται αναφορά στα θύματα του Ισραήλ. Καλά τα είπατε Πρέπει να είναι ε, πρώτο μέλημά μας να προστατεύσουμε τα θύματα της τρομοκρατίας και αυτό θα κάνουμε. Και θέλουμε ε, επίσης να αναπτυχθεί η οδηγία. Πέρα από το χαρτί πρέπει να τους δώσουμε πνοή, ζωή ε, και να πιστέψουμε στα κείμενα των νομοσχεδίων για να, και των οδηγιών για να λειτουργήσουν αισίως και να μας βοηθήσουν στην καθημερινή μας ζωή στην Ευρώπη. Κυρία Ταλή, με ρωτήσατε για τις Βρυξέλλες 2 Ε, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ είμαι ε, δικηγόρος και γνωρίζω πολλούς ε, που πήραν διαζύγιο σε μια χώρα και πρέπει να κινήσουν άλλη διαδικασία για να αναγνωριστεί η απόφαση σε άλλη χώρα. Τι σημαίνει αυτό? Κόστος, γραφειοκρατία, Ε, με αυτές τις Βρυξέλλες 2α η ε, η διαδικασία. Αν έχετε μία απόφαση σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να είναι εκτελεστέα σε οποιοδήποτε άλλο χωρίς να χρειαστεί να περάσει από τον εκτελεστό τίτλο. Εξεκουάτρο το λέμε εμείς οι νομικοί. Αυτό θα ε, κάνει τη διαφορά στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Επίσης, με ρωτήσατε για τα θέματα του Παναμά. Εκπροσωπούμε το Συμβούλιο εδώ. Είμαστε η Προεδρία και όταν μιλώ, μιλώ εξ ονόματος 28 κρατών μελών. Καταλαβαίνετε πώς συζητώ και διαπραγματεύομαι εκπροσωπώντας 28 κράτη-μέλη. Θέλω να ξεκαθαρίσω λοιπόν ότι θα προωθήσουμε τις δύο σχετικές προτάσεις, ποινικοποίηση των αδικημάτων που σχετίζονται με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και αμοιβαία αναγνώριση των εντολών για πάγωμα και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων. Οπότε το πραγματικό ερώτημα είναι, θέλει να πιέσει η Μάλτα για να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή πρόοδο για αυτά τα δύο μέσα, οδηγία και κανονισμός. Ναι, έχουμε αναλάβει αυτή τη δέσμευση. Τι μόνο αυτό. Τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου ε, θέλουμε να την επιτύχουμε μέχρι τον Ιούνιο για την ποινικοποίηση των αδικημάτων που σχετίζονται με την νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων. χθε κάναμε την πρώτη συνάντηση για τι εντολέ επαγώματο και κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων και αυτό είναι έμπρακτη απόδειξη της δέσμευση που έχουμε αναλάβει φυσικά. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα σε άλλες συνθήσεις ε, για την καταπολέμηση φοροδιαφυγής, ε, για ε, το, την νομοποίηση παρανόμων εσόδων. Έχουμε αναλάβει δεσμεύση να σημειωθεί πρώτος για αυτά τα δύο ζητήματα. Επίσης, μιλήσατε για το, το, πρόγραμμα των επενδυτών. Ξαναλέω, εδώ εκπροσωπώ και μιλώ εξ ονόματος 28 κρατών μελών. Δεν μιλώ ως ε, υπουργό της Μάλτας. Σας θυμίζω το Μάρτι. Ε, στις 15 Μαρτίου κάναμε μία σχετική συνάντηση και απαντήσαμε σε όλα τα ερωτήματα και ε, νομίζω διασκεδάσαμε τις ανησυχίες των μελών της Επιτροπής. Μου κάνατε ερωτήσεις επίσης για τη διαφθορά. Και πάλι Δεν εκπροσωπώ μόνο τη χώρα προελευσής μου, αλλά 28 κράτη-μέλη. Και αν μπορούσα να σας πω τι κάναμε για να καταπολεμήσουμε διαφθορά, θα αναφερόμουν ε, σε ένα νομοσχέδιο που κατήργησε την παραγραφή για τα αδικήματα διαφθοράς των πολιτικών. Αυτό ήδη από την αρχή της αιτίας. Αλλά δεν θα μπω, δεν θα αναφερθώ σε αυτά τα νομοσχέδια, διότι δεν είναι ο ρόλος μου εδώ. Εγώ εδώ μιλώ εξ ονόματος των 28 κρατών μελών. Είναι απόλυτη δέσμευση του Συμβουλίου πάντως να σημειωθεί πρόοδος για τα ζητήματα που προανέφερα. Ξαναλέω για την ποινικοποίηση των αδικημάτων σχετίζοντα με την, παρανομ... με την ε, νομοποίηση παρανόμων εσόδων και ε, για το πάγωμα και την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων. Αυτά, γιατί ξεπέρασα για το χρόνο μου και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας. Κύριε Μπονίτσι, πολύ σας ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε που ήρθατε. Καλή τύχη να μου μένει να σας ευχηθώ τώρα. Συνάδελφοι, πρέπει να συνεχίσουμε. θα έρθουν οι συνάδελφοι από την ΕΚΟΝ στις 12 παρατέταρτο. Επόμενο σημείο. Παρουσίαση της πρότασης είπα της του ΟΗΕ για τους ε, ε, πρόσφυγες, για την καλύτερη προστασία των προσφύγων στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο. Με συγκεκριμένες αναφορές στην τρέχουσα κατάσταση στην Ευρώπη. Ε, η ΥΠΑ έχει κάνει πρόσφατα πολύ μεγάλη δουλειά για τις σχέσεις και με τις τρίτες χώρες, με την Τουρκία, παραδείγματο χάρη, ο κ. Κοσετέλ που είναι διευθυντής ε, του, του, μάλλον για την Ευρώπη, ε, θα μας μιλήσει για αυτά που έχουν γίνει στον ΟΗΕ. Σας παρακαλώ, αν έχετε κύριε Κοσετέλ την καλοσύνη, αρχίστε αμέσως. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, που μας ε, προσκάλεσε έτσι ώστε να παρουσιάσουμε κάποιες ε, προτάσεις ε, για την ε, Ευρώπη. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη συνδιαμόρφωση της πολιτικής ασύλου για το μέλλον. Έχετε επανειλημμένα αναφερθεί στην ανάγκη αυξημένης αλληλεγγύης καθώς επίσης και τροποποίησης του Δουβλίνου. Ακούσαμε τις προτεραιότητες της Μάλτας για τους επόμενους έξι μήνες και θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες από τις προτάσεις που κάναμε ε, και στην Μαλτέζικη και στην μελλοντική η Εστονική Προεδρία. Ε, Βεβαίω θα είμαστε και λίγο πιο συγκεκριμένοι, λαμβάνοντα υπόψη και τα όσα ακούσαμε σήμερα το πρωί. Ο κύριο ε, Φίφο Γκράντι στι 5 ε, Δεκεμβρίου τη προηγούμενη χρονιά, ε, εξ ονόματο τη ΥΠΑ τη Αρμοστία, δημοσίευσε κάποιε προτάσει για την προστασία των μεταναστών και των προσφύγων. Αυτές οι προτάσεις είναι συγκεκριμένες και αποσκοπούν στη διαμόρφωση μιας νέας μορφής συνεργασίας που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη αλλά και στα μαθήματα τα οποία διδάχθημεν κατά τα έτη 2015, 2015 και 2016. Ε, σε αυτό το έγγραφο γίνεται αναφορά στην εξωτερική αλληλεγγύη, τα εξωτερικά σύνορα, ε, καθώς επίσης ε, και σε θέματα τα οποία θα αναπτυχθούν περαιτέρω και την 25η Ιανουαρίου. Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ κυρίως στην ανάπτυξη ασφαλών ε, και νομίμων διαδρόμων μέσω των οποίων θα μπορούσαν να φτάσουν οι μετανάστες στην Ευρώπη. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Όταν συζητήσαμε το Migration Compact, ε, καθώς επίσης και τα προγράμματα περιφερειακής προστασίας, ε, συζητήθηκαν και όταν συζητούμε λοιπόν όλα αυτά και τις περιφερειακές και συνεργασίες και συνεργασίες γειτονίας, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούμε και σε αυτούς τους ασφαλείς ε, διαδρόμους. Στο έγγραφό μας ε, αναφέρονται κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, όπως είπα και προηγουμένως, για την αναμόρφωση του συστήματος ε, για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Κάποιες από τις προτάσεις ξεπερνούν και τις προτάσεις που έχει κάνει η Κομισιόν. Έχουμε την αίσθηση ότι μερικές φορές η Κομισιόν δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη ε, τα όσα συμβαίνουν και τα όσα δεν ε, συνέβησαν τα έτη 15 και 16. Ορισμένα σημεία να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα ζητούμε κοινό σύστημα καταχώρησης έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι όσοι φτάνουν στην Ευρώπη καταγράφονται με τον ίδιο τρόπο μέσω του ιδίου συστήματος και ότι τα στοιχεία είναι ε, συνολικά και γνωστά σε όλους ταυτοχρόνως. Αυτό θα βοηθήσει τους ανθρώπους ε, πιο γρήγορα να προωθηθούν στις σωστές ε, διαδικασίες ε, και να καλυφθούν από προστασία όσοι χρήζουν προστασίας και αυτό γρηγορότερα. Ένα τέτοιο σύστημα θα δώσει την αδυνατότητα ανάκτησης εμπιστοσύνης ε, στο σύστημα και θα βελτιώσει τη σχέση με τους ε, πολίτες ε, της Ευρώπης οι οποίοι έχουν τρομοκρατηθεί ενδεχομένως, προβληματιστεί από μη καταγεγραμμένους και καταχωρισμένους πρόσφυγες οι οποίοι κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Ε, επίσης να σας πω ότι υπάρχουν πέντε παράλληλα συστήματα μη συνδεδεμένα μεταξύ τους για την καταχώρηση ε, των εισερχομένων. Ε, αυτό θα βοηθήσει λοιπόν και το screening από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, ε, συγκεκριμένες πρακτικές προτάσεις για τον μηχανισμό καταμερισμού έτσι ώστε να λειτουργήσει σωστά η επανεγκατάσταση γιατί ο αριθμός των επανεγκατεστημένων είναι ε, ε, ιδιαιτέρως ε, και απαράδεκτα χαμηλός. Το θέμα δεν είναι μονάχα θέμα αλληλεγγύης, είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να λυθεί μονάχα από την γεωγραφική κατανομή έτσι όπως συμβαίνει σήμερα. Τρίτη πρόταση Ορισμένοι ε, λένε ότι θα πρέπει κάποιοι ετούντες άσυλο να προχωρήσουν μέσω επισφυρισμένων διαδικασιών, τοχυτέρων διαδικασιών ε, στα σύνορα, έτσι ώστε να προστατευτούν αυτοί που χρειάζονται διεθνή προστασία και να επαναπροωθηθούν αυτοί που δεν έχουν δικαίωμα. Τέταρτον, ε, τα μη ε, συνοδευόμενα παιδιά ε, είναι ένα σημαντικό θέμα. Εμείς πιστεύουμε ότι τα παιδιά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως παιδιά. Πολλές είναι οι συστάσεις και τα νομοθετήματα τα οποία υφίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά λείπει η κοινή πρακτική. Θα πρέπει να σταματήσουμε πλέον να ταχυδακτηλουργούμε όσον αφορά το θέμα αυτό και θα πρέπει γρήγορα να προωθούνται οι διαδικασίες για τον καθορισμό επιμελητών κηδεμόνων είναι πολλές οι περιπτώσεις στις οποίες για διάφορους λόγους δεν υπάρχει δυνατότητα ε, ε, ε, για τον ορισμό κηδεμόνων. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα αναζήτησης των της οικογένειας και των γονέων γιατί αυτό λείπει σήμερα στην Σικελία, στην Ιταλία. Είναι εκατοντάδες τα παιδιά τα οποία φτάνουν ε, με ε, τις ε, βάρκες και το πρώτο ερώτημα είναι υπάρχει δυνατότητα να βρεθούν οι γονείς πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, να γίνει συζήτηση επ' αυτού του θέματος ε, με πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ε, είναι συνήθις και συστηματική διαδικασία η προώθηση των παιδιών στη διαδικασία ασύλου που δεν είναι πάντα προς το συμφέρον τους. Πέμπτον, καλούμε την Ευρώπη να προετοιμαστεί για νέα αύξηση ροών. Ενδεχομένως και ευελπιστούμε ότι δεν θα συμβεί ενδεχομένως δεν θα συμβεί, ωστόσο μας απασχολεί ιδιαίτερος ότι ε, σε σειρά περιπτώσεων φαίνεται η Ευρώπη να μην έχει ούτε πλάν Α ούτε πλάν Β. Κανένα σχέδιο λοιπόν να μην ε, λησμονούμε ότι δεν έχουν ε, σημαντικά τροποποιηθεί οι γενεσιουργές, γενεσιουργές αιτίες των μεταναστών μεταναστευτικών ροών και δεν φαίνεται να απαλληφθούν αυτές οι αιτίες στο μέλλον. είναι πάρα πολύ δύσκολες οι διαδικασίες. Τι να σας πω τώρα, πόσους μήνες ε, χρειαστήκαμε έτσι ώστε να οργανωθούν τα ελληνικά νησιά ε, με, τις, ε, με τα μηχανήματα Eurodac, με τα containers και τα λοιπά. Ξέρουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει οι προσπάθειες να επιταχυνθούν. Έκτο και τελευταίο ακούσαμε ε, πολλά σχόλια παρόμοια στην προηγούμενη συζήτηση για τη Μαλτέζικη Προεδρία, ότι χρειαζόμαστε δηλαδή περισσότερες, περισσότερη επένδυση όσον αφορά την ε, ένταξη ε, των νεοαφιχθέντων. Μέσω αυτής της ένταξης της integration θα, θα αποφευχθούν φαινόμενα αδιαλαξίας, έλλειψης ενοχής και ξενοφοβίας. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των ανθρώπων που φτάνουν και ζητούν τη βοήθεια και βεβαίως ε, θα πρέπει ε, να βεβαιωθούμε ότι γίνονται σεβαστές από όλους οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι θεμελιώδες αρχές. Τέλος, σας ενθαρρύνουμε να δείτε τον τρόπο με τον οποίο ορισμένες από τις προτάσεις αυτές θα μπορούσαν να ενταχθούν ή στην ε, ε, νέα μορφή του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Ιδιαίτερως θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ε, στο γεγονός ότι οι προτάσεις μας για επιταχυμένες διαδικασίες θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τις διαδικασίες καταχώρησης γιατί αυτές οι διαδικασίες για την αποδοχή ή όχι, ε, μας προκαλούν μεγάλες ανησυχίες. Έχουμε δει και τα πράγματα πώς έχουν πάει στην Ελλάδα. Δεύτερον, ε, στην παρούσα συζήτηση μπορούν να συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα, γιατί πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει το 2017 να τα λάβει όλα αυτά υπόψη. Τρίτον, πρότασή μας είναι να υπάρξουν υποχρεωτικές απαιτήσει ότι 30% των ε, πόρων ε, ε, ετησίως ε, να αφορούν την ένταξη. Υπάρχουν χώρες οι οποίες ούτε ένα ευρώ δεν δίνουν για την ένταξη και μετά μας εκπλήσει η κατάσταση στην Ευρώπη και μετά μας εκπλήσει που ορισμένες χώρες στην Ευρώπη δεν έχουν καθόλου πρόσφυγες. Πώς είναι δυνατόν να μην ταπανώνται χρήματα για την ένταξη όλων αυτών των νέων ανθρώπων. Αυτό μας ξεπερνάει έχω χρόνο έτσι ώστε να ασχοληθώ με εξειδικευμένα ζητήματα για την κατάσταση στην Ιταλία, στην Ελλάδα ή στην Τουρκία, αλλά βεβαίως ε, μπορείτε να μου κάνετε ερωτήσεις και θα τις απαντήσω όσον αφορά τις τρέχουσες εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ. Και θα, τώρα θα πάρουν τον λόγο η συνάδελφοι, ο κύριος ε, Λόπες Αγγιγιάρ. Yes. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Κύριε Κοστέλ, εκπροσωπώντας ε, την οπτική γωνία της ΥΠΑ τη Αρμοστίας του Ρέιος Πρόσφυγε. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη δουλειά σα. Πέραν ε, ε, των τεράστιων διαστάσεων αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης, εκτιμούμε το έργο σας ευρύτερα. Θα ήθελα να θίξω κάτι το οποίο με απασχολεί ως εισηγητή του κώδικα θεωρήσεων. Είναι οι ανθρωπιστικές ε, θεωρήσεις. Εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έχουμε κάνει μία σειρά ακροάσεων και συνδιασκέψεων. Και ακούσαμε από πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις, και από εξειδικευμένους ε, ομιλητές και οι δήμονες τη σημασία της διαμόρφωσης νόμιμων οδών που θα διευκολύνουν τα πράγματα για όλους εκείνους που θέλουν να φτάσουν στην Ευρώπη για, ανθρωπιστικούς λόγους. Καθώς ε, διώκονται ε, λόγω ε, θρησκείας, ιδεολογίας κτλ. Λόγω του κοινωνικού του υποβάθρου. Και έτσι υπάρχει ατομικός ή συλλογικός ε, κίνδυνος και απειλή σε συγκεκριμένες ε, ζώνες συγκρούσεων και εμπόλεμες ζώνες. Θα θέλαμε και εμείς λοιπόν ε, να λάβουμε σαφή θέση για το ζήτημα, γιατί ε, ερχόμαστε αντιμέτωποι με σημαντική αντίσταση σε ό,τι αφορά τη χορήγηση ανθρωπιστικών θεωρήσεων στο πλαίσιο του κώδικα θεωρήσεων από τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο. Και θεωρώ ότι μία τέτοια ανοιχτή ε, θέση από την ύπατη ε, αρμοστία του ΙΕ για αλλά και από άλλους οργανισμούς, είναι μια σημαντική κίνηση για να διαμορφωθεί ένα κλίμα που καθώς θα περνάει ο καιρός ε, θα καθιστά σαφές ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτό το φαινόμενο των θαυπιστικών θεωρήσεων στην Ευρώπη. Γιατί αυτό τονίζει την ευθύνη και των κρατών μελών ε, ενώπιον της ανθρωπιστικής ε, τραγωδίας, αλλά και σε αφορά τα νομικά, ε, τους νομικούς κανόνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή από τα θεσμικά όργανα και πιο συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που ακριβώς έχει καταδικάσει το βασίλειο του Βελγίου γιατί αρνείται να τηρήσει την απόφαση που ξεκαθαρίζει την υποχρέωση του Βελγίου να χορηγεί ανθρωπιστικές ε, θεωρήσεις όταν ε, του ζητήθηκε ε, από μία συριακή οικογένεια στο, στην πρεσβεία στο Λίβανο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που κάνετε για τους πρόσφυγες. Διάβασα την ε, πρότασή σας, ε, είναι εύληπτη, όμως ε, παρόλα αυτά έχω διάφορες ερωτήσεις για την καταγραφή αυτά που προτείνεται παραδείγματο χάρη στα hot spot και μετά που περνάμε στο δεύτερο βήμα και βλέπουμε αν έχει ο πρόσφυγας η οικογένεια σε κάποιο άλλο κράτος μέλος το τρίτο βήμα είναι να τον στείλουμε εκεί πέρα που είναι η οικογένεια, οι συγγενείς. Ερώτηση λοιπόν, για να δούμε, να πάρουμε το παράδειγμα της Γερμανίας και της Σουηδίας, ε, που υποδέχτηκαν πάρα πολλούς πρόσφυγες τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουμε τις ποσοστώσεις. Όταν πληρούνται οι ποσοστώσεις λοιπόν, τι θα κάνουμε, θα τους στέλνουμε εκεί ή θα στέλνουμε τους πρόσφυγες σε άλλα κράτη-μέλη. Η Σουηδία ε, ξέρετε, ε, έχει πάρα πολλούς που θέλουν να επανενωθούν οικογενειακά με τους συγγενείς τους, ε, αλλά έχουμε δικούς μας κανόνες ε, για τους συγγενείς. Δεν πρέπει να γίνονται σεβαστές οι εθνικές νομοθεσίες για τα, τη μεταναστευτική πολιτική και την πολιτική ασύλου για να μπορείς να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Δηλαδή, εγώ αναρωτιέμαι για αυτό το βήμα, αυτό που λέτε ότι πρέπει να σταλούν οι πρόσφυγες εκεί που είναι οι συγγενείς τους. Αυτό δημιουργεί προβλήματα με τις ποσοστό. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα, ναι. ε, η κατανομή ε, των ε, ποσοστώσεων. Όταν μιλάμε για τη Λιθουανία και την Ισπανία, που έχουν μικρότερες ποσοστώσεις. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους που δεν θέλουν να πάνε σε αυτές τις χώρες που τους στέλνουμε. Ε, και νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ένα κοινό σύστημα, αλλά πώς θα γίνει να ε, διευκολύνουμε τη διαδικασία με τα κράτη-μέλη που δεν που δεν κάνουν αυτά που πρέπει. Παραδείγματο χάρη στον τομέα της υγείας, δεν έχουν αρκετούς επαγγελματίες. Ε, πώς θα εφαρμοστεί αυτό το κοινό σύστημα. Ευχαριστούμε κυρία Γκόμες. Εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ. κύριε Κοστέλ. για την ε, αυστηρή μεν ε, αξιολόγηση, όμως Πρέπει να τα ακούσουμε όλα αυτά και εμεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα ευχαριστώ και για τι προτάσει σα. Θα ήθελα να μα πείτε μερικά λόγια ακόμα σε ό,τι αφορά τον ε, μηχανισμό κατανομή ε, ε, στα κράτη-μέλη και τι συγκεκριμένε προτάσει σα. Εκτιμώ ιδιαίτερα στις προειδοποιήσεις σας σε ό,τι αφορά τους ανηλίκους. Είναι εξοργιστικό που μιλούμε για ανηλίκους αλλά μιλάμε για παιδιά. Πρέπει να τους μεταχειριζόμαστε ως παιδιά λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε. Ε, σημαντική είναι και η έμφαση που δώσατε στην ένταξη και τον μηχανισμό που προτείνατε, γιατί και αυτό είναι τμήμα του προβλήματος, για να αποφεύγουμε και τις δευτερογενείς μετακινήσεις. Θα ήθελα όμως να μας πείτε πιο συγκεκριμένα και για τον μηχανισμό κατανομής. Βεβαίω έχετε δίκιο ότι ο κατακαιρματισμό που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά την ε, καταγραφή κάτι μη αποτελεσματικό. Και ο Τζόσεφ ασκούσε πιέσεις για την ομάδα ε, Γεζίντη που βρήκαμε στην ε, Ελλάδα. Είχαν καταγραφεί πριν από ένα μήνα και στην Πορτογαλία που είχε δηλώσει ότι θέλει να τους υποδεχθεί, δεν πήγαν ποτέ οι αιτήσει τους. Δεν είχαν ε, ελεγχθεί οι αιτήσει λοιπόν. Εμείς ήμασταν εκεί πριν από ένα μήνα. Και ένα μήνα μετά ακόμα δεν έχουν φτάσει. Είναι εξοργιστική η κατάσταση και είδαμε ότι είχαμε ήδη 600 άτομα από αυτή την κοινότητα των 1.100 ατόμων που είχαν καταγραφεί. Παρά το γεγονό λοιπόν ότι τα 600 αυτά άτομα είχαν καταγραφεί από τα μέσα Δεκεμβρίου, καμία από αυτές τις αιτήσει δεν είχε περάσει τη διαδικασία της ε, επανεκατάσταση. Και αυτό συνδεόταν με το γεγονό ότι η ε, ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες ε, παρουσίασε κάποια ερμηνεία που θα τους έδινε προτεραιότητα. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει θέμα να τους δοθεί προτεραιότητα, παρότι αν ε, συμφωνήσουμε ότι οι γεζίδι είναι θύματα γενοκτονίας, τότε όντως θα πρέπει να λάβουν προτεραιότητα. Σίγουρα όμως δεν τους αξίζει αρνητική διακριτική μεταχείριση. Και αφόσον ήδη είχαν καταγραφεί 600 άτομα, ε, και καμία από τι αιτήσει δεν είχε ε, εξεταστεί, σίγουρα υπήρχε αρνητική διακριτική μεταχείριση. Ποια είναι η θέση τη ΥΠΑ τη Αρμοστία για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε κυρία Γκόμε. Ο κυρίας Βέλτερ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Βρίσκω ο, πάρα πολύ σημαντικά τα στοιχεία που αντλείται από αυτή την ομολογουμένως πολύ δύσκολη κατάσταση. Ε, λέτε ότι πρέπει να υπάρχουν νόμιμοι οδοί μετανάστευσης και συμφωνούμε και άρα πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας ε, σε αυτό. Είναι μια πολύ σημαντική πτυχή της μετανάστευσης. Ε, θα οξυνθούν τα προβλήματα τη, τους επόμενους μήνες. Γιατί πέρα από τα προβλήματα για αυτούς τους ανθρώπους θα έχουμε και προβλήματα ασφαλείας ε, εάν δεν καταφέρουμε να αποτρέψουμε και να αναχαιτήσουμε αυτές τις, τις τάσεις. Ε, ε πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ε, χειραγωγείται αυτό το θέμα, υπάρχει προπαγάνδα και ε, το εκμεταλλεύονται κάποιοι, ε, αλλά το σύστημα καταγραφής είναι σκανδαλώδες που χρειάζονται μήνες ολόκληροι για να καταγραφούν αυτά τα δεδομένα. Χρειάζεται ίσως ένα σύστημα προεγγραφής ε, και μας είπαν κάποιοι πρόσφυγες, ε, μας ε, κατέγραψαν τον Απρίλιο, δηλαδή είναι σε αυτή την φάση προεγγραφής 8 μήνες οι άνθρωποι, μα είναι παράλογο αυτό. Και αν δεν κάνουμε κάτι για να σώσουμε την κατάσταση με τη γραφειοκρατία δεν θα επιτύχουμε τίποτα. Οι τραγικές εικόνες από την Ελλάδα τώρα. Ε, έτυχε να είναι ιδιαίτερα βαρύς ε, ο χειμώνας ε, φέτος. Ε, υπήρχαν προειδοποιήσεις και βλέπουμε όμως ότι ε, κολλάνε τα πράγματα στη γραφειοκρατία. Πρέπει λοιπόν να απομακρυνθούμε από αυτές τις διατάξεις. Έχουμε αυτό το case name και κολλάει η διαδικασία. Ε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι ενδεχομένως η λύση είναι να είναι πιο ευέλικτο το σύστημα, είναι κάποιοι που μπορούν να πάνε σε άλλες χώρες, άλλοι που δεν μπορούν, είναι χαοτικό το σύστημα και ε, χρειάζεται μια ομάδα εργασίας, πιστεύω. Πρέπει ρεαλιστικά και ταχύτατα να ε, επεξεργαστούμε αυτούς τους φακέλους, ε, γιατί το θέμα είναι ανθρώπινες ζωές, όπως είπε και η κυρία Γκόμες. Όταν ε, πολλούν τις γυναίκες και είναι ε, ε, κρατούνται από τον ίσης τόσους μήνες και μετά περιμένουν 8 μήνες μέχρι τον Απρίλιο για να επεξεργαστούμε εμείς την αίτησή του. καταλαβαίνετε ε, πόσο παράλογο είναι αυτό το σύστημα. Ευχαριστώ, Βίξτρομ. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Θα διαβάζω το έγγραφο, αυτό το, αυτή την προσούρα που μας δώσατε και πραγματικά πιστεύω ότι ε, μας βοηθάτε πολύ στην μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι ένα έγγραφο το οποίο ακριβώς αναφέρεται σε αυτά που πρέπει να κάνουμε πιστεύουμε ότι θα, αυτά τα θέματα της εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων, της αλληλεγγύης είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα ήθελα ε, να ξέρω, γιατί ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει η εργασία γι' αυτό και προσπαθούμε τώρα να ε, ε, δημιουργήσουμε ένα ανθεκτικό, ένα ισχυρό σύστημα, ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου <clears throat> και να ξαναδούμε το θέμα του Δουβλίνου. Ε, και γνωρίζουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί πολλές ε, χώρες ε, έχουν ιδιαίτερα αρνητική στάση ακόμα και στο να συνεργαστούν και να συζητήσουν. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα σύστημα βάση ποσοστώσεων. Εν πάση περιπτώσει όμως εγώ θα ήθελα ε, να ασχοληθώ λίγο με το θέμα του Δουβλίνου έτσι όπως ε, προωθείται από την Κομισιόν γιατί βλέπω ε, εδώ τις προτάσεις σας και πραγματικά κουμπώνει πάρα πολύ καλά με αυτά που θα θέλαμε εμείς. Μιλάμε για τον κανονισμό του Λονδίνου, μιλάμε για άλλα νομοθετικά εργαλεία επί των οποίων εργαζόμαστε και θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό που υπόθηκε και προηγουμένως, ε, γιατί ακριβώς εκεί έγκυται ε, μία από τις δυσκολίες ε, της νέας πρότασης Δουβλίνου. Πώς θα αντιμετωπίσουμε δηλαδή και πώς θα προστατέψουμε τους ασυνόδευτους ανήλικους. Ξέρουμε ότι πέρσι τουλάχιστον 10.000 νέοι παιδιά και έφηβοι εξαφανίστηκαν, τους χάσαμε. Ε, και ξέρουμε ότι υφίστανται ε, ε, προβλήματα και κακοποιούνται τα παιδιά αυτά όχι στην Ευρώπη μόνο αλλά και σε όλο τον κόσμο. Επομένω θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι θα κάνουμε τα παιδιά αυτά. Όσον αφορά τώρα την ένταξη ε, στην κοινωνία. Μετά από την διάσκεψη ε, του Σεπτεμβρίου ε, η ένταξη βρίσκεται πλέον, έχει βρει τη θέση της στις δηλώσεις του Συμβουλίου. Οι κυβερνήσεις, οι αρχές θα πρέπει πλέον να ε, ε, έχουν ε, την ευθύνη για τα θέματα αυτά, αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα και τα πανεπιστήμια και τα σχολιά και όλοι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όμως ξέρετε ότι αυτό είναι εθνική αρμοδιότητα. Ωστόσο έχουμε κάποια καλά παραδείγματα τα οποία μπορούμε να μοιραστούμε με άλλους, αλλά θα μπορούσατε να επιστρέψετε στις πραγματικές συγκεκριμένες απτές προτάσεις όσον αφορά την υποχρεωτική το υποχρεωτικό μοίρασμα ευθυνών ε, υπό το Δουβλίνο και στο κοινό σύστημα καταγραφής. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Σλάιμα. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με την συνάδελφο Σισίλια Βέλστρομ ότι είναι πολύ επίκαιρη η παρουσίασή σας και εγώ βεβαίως εκτιμώ πολύ τις προσπάθειες που καταβάλλετε έτσι ώστε ε, να βρείτε κάποιες ε, εναλλακτικές ε, λύσεις σε σχέση με την μεγάλη προτεραιότητα της οικογενειακής επανένωσης αλλά και της ευρύτερης οικογενειακής επανένωσης. Και μας μας απασχολεί αυτό πολύ. Το ε, ζήτημα είναι τι προτείνει η μεταρρύθμιση της ε, πρότασης ε, για το Δουβλίνο στο σημείο 3, δάφιο 3 και αυτό το λεγόμενο inadmissibility check Ε, πρόκειται για μία ε, έννοια η οποία ε, δεν αποτελεί ευρωπαϊκή έννοια και είναι άλλωστε και μία έννοια που δεν βοηθάει την προώθηση της συζήτησης για τον ευρωπαϊκό κατάλογο των ασφαλών χωρών ε, η πρώτη χώρα εισδοχής ε, είναι αυτή η οποία θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσον ε, είναι αποδεκτή, αποδεκτό ή όχι το αίτημα βάσει της αρχής της ασφαλούς χώρας ή εναλλακτικά θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη αντίδραση για, την, για το συγκεκριμένο αίτημα ασύλου. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί όμως ένα φίλτρο το οποίο θα μπορεί να φτάσει στο 70-80% Αναφέρομαι τώρα στη χώρα μου στην Ιταλία. Τι θα γίνει εάν ε, ε, και κάποιες άλλες ε, χώρες θεωρούνται πιο ασφαλής χώρα. Ας πούμε το Αφγανιστάν να θεωρείται πιο ασφαλής χώρα γιατί είδαμε ότι υπάρχουν κάποιες εξελίξεις σε σχέση με το Αφγανιστάν. Έχετε μήπως και εσείς την αίσθηση ότι αυτό το inadmissibility check, το 3, παράγραφος 3 μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ε, πριν ακόμα ε, ε, ληφθεί υπόψη το κατά πόσον ο νεοεισερχόμενος είναι ανήλικας, έχει ανάγκη τα κτλ. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Ο προβληματισμός είναι ο εξής. Βλέπω ότι υπάρχει αυτή η πρόταση για ε, περιπτώσεις ε, ε, προδήλως αβάσιμες βάσει της πρώτης διαδικασίας στην χώρα εισόδου. Αλλά αυτό με προβληματίζει λίγο γιατί ξέρετε είναι πολύ βαριές οι διαδικασίες αυτές. Είναι πολύ βαριέ και περίπλοκες οι διαδικασίες αυτές ε, όσον αφορά ε, τα αιτήματα ασύλου. Όσον αφορά τώρα τα ελληνικά νησιά, ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βοηθηθούν να φύγουν οι άνθρωποι αυτοί από τα νησιά και να σταλούν στην ενδοχώρα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί η κατάσταση είναι τραγική. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον εκπρόσωπο τη ΥΠΑ τη για τη δουλειά που κάνουν και για τη συνεργασία μαζί μα Εγώ είμαι η για την πρόταση για το πρόγραμμα επιστροφών ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ που τονίσατε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε νόμιμες οδούς μετανάστευσης. Ε, πρέπει να υπάρχουν ε, διαφορετικοί τρόποι, ανθρωπιστική θεώρηση, οικογενειακή επανένωση κτλ. Ε, για τις επιστροφές, ε, συνεργαζόμαστε στενά και ε, εγώ βασίζομαι στο ότι το μοντέλο τη, της ΥΠΑ της θα πρέπει να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για μας. Ε, υπάρχουν διάφορες ελλείψεις μέσα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεργαζόμαστε εδώ με τα μέλη της Επιτροπής για να προτείνουμε αναβάθμιση αυτής της πρότασης. Ε, σίγουρα θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι σχέση με τον αριθμό των προσφύγων. Ε, σίγουρα πρέπει να βοηθήσουμε πολύ περισσότερους ανθρώπου. Εκατοντάδε χιλιάδε. το άρθρο 4 είναι ιδιαίτερα προβληματικό διότι εκεί εντάσσεται η Συμφωνία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ε, και Ε, και αποκλίνουμε έτσι από το πρότυπο της ε, είπα τις αρμοστίας και ήθελα την ε, άποψή σας γιατί όπως σας είπα προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βοηθήσουμε καλύτερα τους πρόσφυγες και να βρούμε περισσότερες νόμιμες οδούς μετανάστευσης και κάτι άλλο τώρα σε σχέση με τη δική σας πρόταση ε, δεν θα σταθώ στα θετικά σημεία για τους ανήλικους και το καθεξής. Αυτή οι ε, ε, σπευσμένη συνοριακή έλεγχη μα ανησυχούν λίγο. Ε, είπε και η Ιταλίδα συνάδελφος και έχει δίκιο για να είναι για να λειτουργήσει εύρυθμα το σύστημα θα πρέπει να αυξηθούν οι Ε, να αυξηθούν οι απελάσεις ε, και δεν ξέρω ε, πώς ακριβώς μπορούμε να βρούμε μια άλλη λύση. Στην Ελλάδα είναι τραγική η κατάσταση. Λέμε ότι δεν πρέπει να υιοθετήσουμε το αυστραλιανό σύστημα και να το στέλνουμε σε μακρινά νησιά, αλλά τελικά αυτό κάνουμε. Για να μην τους βλέπουμε θα πρέπει να κάνουμε κάτι αμελητή και θα ήθελα να ενθαρρύνω και τους συναδέλφους να πιέσουν. Ναι, τελειώνω, Πρόεδρε. Η Μαλτέζικη Προεδρία μας είπε ότι θα πρέπει όχι μόνο να συνεχίσουμε να εφαρμόσουμε τη συμφωνία με την Τουρκία, να φτιάξουμε και καινούργια με τη Λιβύη. Και θέλω να μου πείτε εσείς τι πιστεύετε. Ευχαριστούμε. Έχουμε άλλους τέσσερις ομιλητές που θέλουν να παρέμβουν. Ε. Νομίζω ενδιαφέρεστε όλοι και για τις απαντήσεις. Ε, στις 11 στις 12 ε, παρατέταρτο αρχίζει η κοινή συνεδρίαση. Ε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι συνεργάσιμη. Θα ήθελα να καταλάβω ποια είναι η άποψη τη ΥΠΑ τη Αρμοστία και του πρόσφυγε, σε ό,τι αφορά την ε, πρόταση επανεγκατάσταση. Ε, ήδη η κυρία Βιόρκα αναφέρθηκε. Θεωρείτε ότι η επανεγκατάσταση θα αυξηθεί στην Ευρώπη. Γιατί εγώ πολύ αμφιβάλλω. Θα ήθελα όμως να δω τη δική σας ε, γνώμη, γιατί τα στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ χαμηλά. Φαντάζομαι ότι επαγνωσμένα θέλετε να αυξηθούν αυτό είναι το μέσο που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Σαρτζεντίνη. Κυρία Κέγγε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω κι εγώ να είμαι σύντομη. με μεγάλη χαρά άκουσα τα όσα είχατε να μας πείτε, ε, κυρίως όσον αφορά το κοινό σύστημα, το κοινό διοικητικό σύστημα ε, και το, συνθήκε συνθήκες υποδοχής ε, και ένταξης. Ε, αλλά για να τα καταφέρουμε αυτά θα πρέπει οπωσδήποτε ε, πρώτα να έχουμε μία διοικητική απλούστευση. Πριν δηλαδή τους υποδεχθούμε και τους εντάξουμε θα πρέπει να τους καταγράψουμε. Δυστυχώς όμως ε, η γραφειοκρατία είναι μακρά και επομένως δεν διευκολύνεται η υποδοχή των ανθρώπων. Σε χώρες όπου, όπως η Ιταλία και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα. Η Ιταλία πάντως έχει προωθήσει ε, μια καλή πρόταση για την ε, υποδοχή, αλλά δυστυχώς ε, η έλλειψη ελληνικής δεν βοηθάει. Ερώτηση. Για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την επίγουσα κατάσταση και την υποδοχή σε αυτά τα μεγάλα κέντρα, ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις σας εγώ θα ήθελα μία διασπαρμένη υποδοχή σε ολόκληρη την επικράτεια. Συμφωνείτε με αυτό. Ma Vorrei esprimere la mia gratitudine. Θα ήθελα ε, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την ύπατη ε, για τους πρόσφυγες ε, σε σχέση με τις προτάσεις που έχει υποβάλει με μία φράση που είπατε και που αναφέρεται εδώ με εντυπωσίασε ιδιαιτέρως εάν δεν δημιουργήσουμε ασφαλείς διαδρόμους προς την Ευρώπη τότε θα δημιουργήσουμε μία τεράστια underclass και πραγματικά ε, αυτή είναι μια πολύ ξεκάθαρη θέση της ΥΠΑ της Αρμοστίας όσον αφορά την ε, Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας διότι είναι μια ε, συμφωνία, πώς να σας το πω, η οποία μπάζει από κάθε πλευρά. Δεν είναι μοντέλο ε, ε, σωστό, ωστόσο είναι ένα μοντέλο το οποίο αντιγράφεται πλέον ε, και στη συμφωνία με τη Λιβύη, χώρα ιδιαιτέρως ασταθεί Υπάρχουν πολεμικά πλοία Ιταλικά στα χωρικά ύδατα της Λιβύης και τι να σας πω τώρα, εγώ δεν καταλαβαίνω πώς ε, μπορεί να αποτελέσει πρότυπο η συμφωνία με την Τουρκία τη στιγμή που έχουμε εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στα ελληνικά νησιά. Και παρόλα αυτά, και παρόλα αυτά συνεχίζουμε να λέμε ότι οι πρόσφυγες ε, που έφτασαν στην ε, Ελλάδα και μετά στην, Ελλάδα, στην ε, Ευρώπη θα πρέπει να ξαναγυρίσουν στην ε, Ελλάδα και ότι είναι εξαιρετική η συμφωνία με την Τουρκία παρά τις παραβιάσεις οι οποίες γνωρίζουμε ότι λαμβάνουν χώρα στην Τουρκία. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πώς είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι είναι πρότυπο η συμφωνία αυτή και θέλω να μου πείτε την άποψή σας γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα είμαι σύντομη λέει η κυρία Χιμένες. Ε, με απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα του τράφικινγκ, διακίνησης ε, ε, ανθρωπίνων όντων. Με απασχολεί ιδιαίτερα, γιατί γνωρίζουμε ότι υφίσταται και στα πλαίσια των προσφύγων και των προσφυγικών ροών. Πώς, μπορείτε, πώς νομίζετε ότι μπορούμε να καταπολεμήσουμε το θέμα αυτό γιατί, γιατί δεν τιμωρείται αναλόγως ε, ε, η διακίνηση ε, ανθρωπίνων όντων, νεαρών, παιδιών, νέων ανθρώπων, γυναικών και η εκμετάλλευσή τους. Αναφερθήκατε στους ασφαλείς διαδρόμους. Μήπως όμως είναι απλά λόγια, Πώς είναι δυνατόν να εφαρμοστούν ε, αυτά λαμβάνοντας υπόψη τις ε, προσφυγικές ε, ροές, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι να υλοποιηθούν πραγματικά λαμβάνοντας υπόψη το εύρος του προβλήματος. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε πολύ δύσκολο έργο να απαντήσετε σε, αυτά τα, σε αυτές τις ερωτήσεις και μάλιστα σε μικρό χρονικό διάστημα. Παρακαλώ λοιπόν παρόλα αυτά να είστε σύντομος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι επικίνδυνη αποστολή ας πούμε. Γι' αυτό καλό θα ήταν να έρθουμε διμερώς και σε επαφή ε, για να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες ε, σε ό,τι αφορά το σύστημα κατανομής, ε, την ανταλλαγή προφοριών με την Επιτροπή που παρουσιάζει προβλήματα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση μέσα σε 7 λεπτά να καταφέρω να απαντήσω σε όλα αυτά. Πρώτον, για τι ανθρωπιστικέ θεωρήσει. Ε, συμφωνούμε απολύτως και το υποστηρίζουμε. Το πρόβλημα είναι ότι ε, κάποιες ε, χώρες αναφέρουν ότι θέλουν να, το, να προχωρήσουν σε αυτό το βήμα, αλλά με το που αναφέρουν αυτή την πρόθεσή τους κατευθείαν κατακλείζονται από αιτήσει. Επομένω, πρέπει να υπάρχει και ένας, ε, μια δικλείδα ασφαλεία, ένα μηχανισμό. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το να έχουμε μια θεώρηση για οικογενειακή επανένωση είναι αδύνατον. Ένα νέο Ερυθρέο ε, που ε, δεν μπορεί να πάρει ε, θεώρηση, να πάει, δεν μπορεί να πάει στο χαρτούμ, δεν μπορεί να πάρει πρόσβαση, δεν έχει πρόσβαση σε διερμηνέα. Δεν έχουμε λοιπόν τα, τα βασικά του ευρωπαϊκού κεκτημένου για αυτούς τους ανθρώπους. Συμφωνούμε όλοι να καταπολεμήσουμε τους ε, διακινητές, να φτιάξουμε ένα σύστημα ασύλου, διαχείρισης, μετανάστευσης στις χώρες διέλευσης, χώρες προέλευσης. Όλοι συμφωνούμε σε αυτά. Αλλά ποια είναι η εναλλακτική για όσους χρήζουν ε, διεθνούς προστασίας. Λείπουν. Δεν υπάρχουν καθόλου σε αυτές τις ε, διμερείς συμφωνίες με κάποιες αυτές τις βασικές χώρες οικογενειακή επανένωση. Γιατί την ιεραρχούμε τώρα ως Γιατί έτσι έχει η πραγματικότητα στην Ευρώπη. Και πάλι χρησιμοποιώ το παράδειγμα του νέου Ερυθρέου που φτάνει στην Ιταλία αυτή τη στιγμή. Ε, έχουμε δύο επιλογές πολιτικά. Είτε του επιτρέπουμε νομίμως να πάει εκεί που είναι η οικογένειά του στην Ευρώπη, είτε παράνομα. Αλλά θα μετακινηθεί το άτομο, ούτως ή άλλως. Ας ασφαλίσουμε, λοιπόν ότι οι ευρωπαϊκοί νόμοι θα λαμβάνουν υπόψη και αυτή η δυναμική που προκύπτει από τους οικογενειακούς δεσμούς. Επομένω, είτε θα το ρυθμίσουμε με το νομικό μας πλαίσιο ε, για να διαμορφώσουμε ένα, μια οδό ασφαλείας, αντί ε, να λέμε ότι δεν θα γίνει ποτέ. Αλλά μην παριστάνουμε ότι δεν θα γίνει ποτέ. Μετά από εκεί πέρα, αν δεν υπάρχουν οι δικλείδες, ε, ναι, όντω θα λέμε ότι δεν υπάρχει το δικαίωμα στην ε, επανεκατάσταση, ότι είναι ένα, ένα μέσο αλληλεγγύης. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες τη φορά το inadmissibility procedure. Ε, βέβαια, χρειάζονται και οι ε, διαδικασίες, αλλά εγώ τα ξέρω εκ των έσω. Αν πάτε στα ελληνικά νησιά, γνωρίζετε έναν επίκο, Μπαγκλαντέ, την Ισία, έναν γεζίδι από το Ιράκ, δεν ε, χρειάζεται μία ώρα για να καταλάβει κανείς αν χρήζει αυτό το άτομο ε, διεθνούς προστασίας ή όχι. Δεν είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα. Ναι, πρόκειται για εφαρμογή του νόμου, αλλά και γνώση της κατάστασης ε, της χώρας προέλευσης. Δεν είναι λοιπόν πυρηνική φυσική, είναι κάτι το οποίο γίνεται πρακτικά. Αυτό θέλουμε να πούμε με αυτή την πρόταση είναι διαχειρίσιμο. 60-70% των ε, περιπτώσεων των ατόμων που καταφτάνουν στην Ευρώπη θα μπορούσαν ε, να του διαχειριστούμε μέσω τη ταχεία διαδικασία. Οι υπόλοιποι μπορούν να πάνε στην ε, κανονική συνήθεια διαδικασία, ιδίω ό,τι αφορά την αξιολόγηση αξιοπιστία. Ασυνόδευτοι ανήλικοι. Ουσιαστικά το συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Δεν θα πρέπει να υποθέτουμε ότι το παιδί χρειάζεται άσυλο, χρειάζεται προστασία Όμω συνήθω η καλύτερη προστασία είναι αυτή που του παρέχει η οικογένειά του, όπου αυτό είναι δυνατόν. αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένα σύστημα το οποίο να προσπαθεί να το επανενώσει το παιδί με την οικογένειά του. Ενσωμάτωση. Είπατε πολλά και σωστά πράγματα. Κάτι το οποίο αναφέρεται στο, στην έκθεσή μας. 30% λέμε των ε, ε, στρατιωτικών δαπανών θα πρέπει να δαπανώνται σε αυτά τα άτομα. όχι όλα αυτά τα χρήματα όμως θα πρέπει να πηγαίνουν στα κράτη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην κοινωνία των πολιτών, κοινέ, ε, τοπικές αρχές. Αυτοί είναι οι φορείς ενσωμάτωσης στην Ευρώπη. Δεν είναι οι κρατικές πολιτικές μόνες. Τα κράτη είναι αυτά που ορίζουν την πολιτική, αλλά από εκεί και πέρα υλοποιείται και σε άλλα επίπεδα. Όχι λοιπόν στο κράτος η χρηματοδότηση, αλλά σε αυτούς τους φορείς. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία δεν μπορεί να ακολουθηθεί και στην περίπτωση τη Λιβύα. Δεν υπάρχει κυβέρνηση αρχικά. Δεν τίθεται ζήτημα. Μετά πρέπει να γίνει και ανάντι μια δουλειά. Όπω είπα και για την Ιταλία. Μόνο 39% των ατόμων που φτάνουν στην Ιταλία. Από του 170.000 άτομα λοιπόν που έχουν φτάσει, 39% ε, χρήζουν προστασία. Οι υπόλοιποι όχι. Πρέπει λοιπόν να επιστραφούν αυτά τα άτομα στη χώρα τους. Πρέπει λοιπόν να τα εξετάσουμε και αυτά. Δεν έχω χρόνο να εξετάσω άλλες στοιχές για την επανακατάσταση. Δεν υπάρχει Ε, αρμοδιότητα του δικού μας φορέα για το ζήτημα αυτό. Είναι θέμα του ΕΑΖΟ. Τώρα, γιατί δεν ε, κινούνται αρκετά γρήγορα το θέμα με τον Γεζίτη. Γιατί κάποιοι είναι ρακινοί και έτσι εξαιρούνται ε, από ε, από το καθεστώς αυτό. Πέφτουν κάτω από το 55% του ε, ποσοστού της το οποίο είναι γελίο. Άλλοι δεν περνούν από το ελληνικό σύστημα ε, αξιολόγησης. Δεν κατανοώ γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Μετά, δεν θα έπρεπε να καταγραφούν στο hotspot αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό δεν έχετε εγκρίνει. Γιατί πρέπει να επανακαταγραφούν δεύτερη φορά λοιπόν. Ή με ρωτάτε, δεν ξέρω. Και πάλι, αυτά άτομα θα τα πράγματα μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε πολύ καλύτερα. Όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ιταλία, ούτε στη Βουλγαρία. Γενικά, αυτές οι προκλήσεις είναι διαχειρίσιμες και θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Δεν έχει χαθεί η μάχη, αλλά πρέπει να τα πάμε καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, απαντήσεις σας. Ε, σίγουρα και μεμονωμένα μπορεί να σας βρει κάποιος για να συνεχίσετε τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε καθυστερήσει λίγο. Ας περάσουμε λοιπόν στην κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΕΚΟΝ σε ό,τι αφορά... Συγγνώμη, όσοι θέλουν να αποχωρήσουν ήσυχα για να προχωρήσουμε κι εμείς. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την πρόληψη χρήση των ε, δημοσιονομικών συστημάτων για, την, ε, για το ξέπλυμα ε, χρήματο για τη χρηματοδότηση τη δημοκρατία. Παρακαλώ, θέλουν να αποχωρήσουν, να το πράξουν ήσυχα για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας.